excellent good morning to all of uh, you. Καλημέρα σε όλους. Ε, και ορίσατε όσοι τώρα φτάσατε στην Επιτροπή μας ε, των Γυναικών τελείωσε η κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξης και τώρα έχουμε το πρώτο σημείο στην ημερήσια μας διάταξη όπου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας ομιλητές αυτή τη στιγμή. Προσβλέπουμε πολύ στη συνεργασία που έχουμε μπροστά μας ε, Καλημέρα στην κυρία Ντάκμαρ Σουμάχερ που είναι ε, ε, αρμόδια διευθύντρια του Γραφείου για τις Γυναίκες του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες, ε, τον πρέσβη Μαουρίσιο Εσκανέρο, επικεφαλής της αποστολής του Μεξικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον πρέσβη Μάρα Μαρινάκη, κύρια σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φύλλο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ε, το σημείο 8 λοιπόν είμαστε στην ημερήσια διάταξη και αφορά το Φόρεμ Ισότητας των Γενεών που είναι μια και μια συγκέντρωση ε, πολιτών που έχει συγκληθεί από τον UN Women και το ε, φιλοξενούν ο διοικητής του Μεξικού και της Γαλλίας. Και εμείς ορισμένοι από εμά ε, σε διμερή βάση είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Είδαμε ότι υπάρχουν Υπάρχει τόσο πολύ ενέργεια και όρεξη για την επερχόμενη αυτή διάσκεψη, φόρουμ, όπου ε, πραγματικά προσβλέπουμε σε αυτό. Θα γίνει στο πόλη ε, του Μεξικού και θα, το αποκορύφωμα θα είναι στο Παρίσι στις 7 και με 10 Ιουλίου. Έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές που θα μας πούν τα πάντα για αυτή την εκδήλωση και πώς θα μπορούσαμε στενά να συνεργαστούμε με τους ε, εμείς οι ευρωβουλευτές μαζί σας. Θα δώσω λοιπόν το λόγο αμέσως στην Τάγμαρ Σουμάχερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία. Είμαι μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ μαζί με το πρέσβη του Μεξικού του Μεξικού και τον πρέσβη της Γαλλίας και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Είναι, σας ευχαριστώ που συγκαλέσατε αυτή τη συνεδρίαση. Προετοιμαζόμαστε το 2019 για το 2020. Είναι μια καλή ευκαιρία ώστε πραγματικά να ε, ανακοινήσουμε τον κόσμο όσον αφορά την ισότητα των φύλων και να συγκεντρώσουμε στήριξη. Θα ήθελα να σας δώσω το πλαίσιο για το φόρουμ ε, για τις γενναίες. Ε, το 2020 είναι πολύ σημαντικό ε, για πολλούς λόγους. 70η επέτειο στο ΟΗΕ, πέντε χρόνια μετά από τους βιώσιμους ε, στόχους, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, έχουμε ε, τη, ε, ψήφισμα 1325 για τις γυναίκες και τα παιδιά και τα δικαιώματά τους και το 2009 επίσης είναι η 40η επέτειος του ΣΥΝΤΟΡ που είναι ε, πολύ σημαντική ε, πέτειος για την ε, προάσπιση και την προαγωγή της ισότητας των φύλων. τώρα, το Φόρουμ Ισότητας των Γενεών, γιατί υπάρχει, για διά, πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι να συγκεντρωθεί και να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών αλλά και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι φορείς Ε, κυβερνήσεις, ιδιωτικό τομέα, ε, τομέας, ε, πανεπιστημιακή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όλοι, είναι το κοινό. Ε, πρέπει πραγματικά να κινητοποιήσουμε τους πάντες ώστε να δημιουργηθεί ένα κίνημα το οποίο πραγματικά να σημάνει τη διαφορά για την ισότητα των φύλων. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε δει μια οπισθοδρόμηση όσον αφορά την ισότητα των φύλων και ο Γενικός μας γραμματέα είπε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε και να αντιστρέψουμε την ατζέντα για την ισότητα των φύλων. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι ως UN γυναίκες που συγκαλούμε εμείς αυτό το φόρουμ και το φιλοξενούμε μαζί με την κυβέρνηση του Μεξικού όπως είπε η ε, πρόεδρος 7 ε, με 10 Μαΐου και μετά με την γαλλική κυβέρνηση από τις 7 μέχρι τις 10 Ιουλίου στο Παρίσι. Είμαστε πολύ ευγνώμονες, σας ευχαριστούμε πολύ και εκτιμούμε ιδιαίτερα την υποστήριξη γιατί και πιστεύουμε πως είναι μια, ένας σπουδαίος συνδυασμός προσπαθειών για τον τρόπο τώρα με τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε. Όπως σας είπα, πρόκειται για μια πορεία που ξεκινά ήδη φέτος. Έχουμε λάβει πολλές εθνικές αναφορές, πάνω από 160 από κυβερνήσεις ολόκληρο τον κόσμο, για το τι έχουν επιτύχει σε σχέση με την ε, πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου που εγκρίθηκε πριν από 25 χρόνια. Ε, Ε, έχουμε, βλέπουμε τι έχει επιτευχθεί, αλλά και πού υπάρχουν ακόμα και να... Ε, εμείς μελετάμε και αναλύουμε αυτές τις εθνικές αναφορές, αλλά και γίνονται και τοπικές διαβουλεύσεις. Ε, έχουμε ολοκληρώσει την περιφερειακή διαβούλευση της Ασίας, είναι υπό εξέλιξη, μάλλον τελείωσε και της Ευρώπης η Ευρωπαϊκή Διαβούλευση ε, είναι πολύ σημαντική η διαδικασία και μετά αυτά όλα τροφοδοτούν την έκθεση του Γενικού Γραμματέα που θα παρουσιαστεί νωρίς του χρόνου και που θα ε, στηριχθούν οι συζητήσεις για την κατάσταση των γυναικών που θα αρχίσουν από τις 9 Μαρτίου. Πολύ ευτυχής είμαι που θα έχουμε εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βεβαίως μπορούμε να βασιστούμε στην ισχυρή παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο CSW. Ε, του χρόνου ε, δεν θα καταλήξουμε σε συμπεφωνημένα συμπεράσματα, αλλά θα έχουμε πολιτική δήλωση που θα εγκριθεί την πρώτη μέρα του CSW και θα έχουμε και μια επαιτειακή συνεδρίαση την ίδια μέρα. Ελπίζουμε να έχουμε υψηλή εκπροσώπηση σε υπουργικό επίπεδο και προσβλέπουμε <clears throat> σε μια ιδιαίτερα ισχύρη ε, ε, σύσκεψη του CSW. Και μετά πάμε στις 7 και 8 Μαΐου στο Μεξικό και ξέρω ότι ο πρέσβης θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για εκεί και αυτό θα σημάνει την έναρξη του Φόρουμ για την Ισότητα των Γενεών. και όπως σας είπα το αποκορύφωμα θα είναι στο Παρίσι τον Ιούλιο. Ποια θα είναι τα πορίσματα, το αποτέλεσμα. Πρόκειται για δημιουργία κινήματος, θέλουμε να συγκεντρώσουμε την κοινωνία των πολιτών, τους νέους και εγώ θέλω να σας πω μια ιστορία. Πολλές Έχω παρακολουθήσει πολλές εκδηλώσεις τους τελευταίους μήνες και όταν ρώτησα το τους νέους αν ξέρουν την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, πολλοί εξ αυτών δεν τη γνωρίζουν ενώ τα θέματα που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου είναι πολύ σημαντικά για τους νέους, αλλά δεν είναι απαραίτητο γνωστό αυτό το έγγραφο. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν με το Φόρουμ Ισότητας των Γενεών είναι ακριβώς να ε, τους φέρουμε κοντά, να ενημερωθούν και να δημιουργήσουμε και συνασπισμούς δράσης. Ε, μπορεί να είναι συνασπισμοί μεταξύ πολλών κρατών που θα συμπεριλαμβάνουν δεσμεύσεις για την ισότητα των φύλων, δεσμεύσεις από κυβερνήσεις, από την κοινωνία των πολιτών, από τον ιδιωτικό τομέα και άλλους φορείς. Αυτό το οποίο Επιθυμούμε είναι οποιοδήποτε θέλει να είναι μέρος μιας τέτοιας, ενός τέτοιου συνασπισμού δράσης και να αντιμετωπιστεί το κενό, το χάσμα που βλέπουμε μεταξύ των γενεών και της ισότητας αυτών. Ε, θέλουμε να έχουμε να αποτελείται από κάποιο κυβέρνηση, δηλαδή η κυβέρνηση που θα εκπροσωπείται από υψηλό επίπεδο, επικεφαλής κράτους δηλαδή και η κυβέρνηση. Δεύτερον, θα πρέπει να δεσμευτεί για τη δράση την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και τρίτον οικονομική δέσμευση για να αντιμετωπίσουν τα θέματα <clears throat> των, ε, της ισότητας των γενναίων. Για την, την ατζέντα θα την ενημερώνουμε τακτικά, οπότε παρακαλώ παρακολουθήστε εκεί τι γίνεται και να αναφέρω ε, γιατί έχουμε βέβαια το Μεξικό και τη Γαλλία, αλλά επίσης θα διοργανώσουμε δορυφορικές συνόδες ώστε να κινητοποιήσουμε και άλλες χώρες και να είναι πραγματικά παγκόσμια η προσπάθεια. Αυτά έχω να σας πω για την ώρα. Προσβλέπω στη συζήτηση που θα κάνουμε. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για το ξεκίνημα του διαλόγου. Τους επόμενους μήνες θα πρέπει να είμαστε πολύ στενή επαφή, να δριάζουμε τακτικά και στο πλαίσιο του CSW, ώστε αυτό το φόρουμ, όπως είπε και η πρόεδρος τόσο όμορφα, να είναι μια πραγματική ειδική στιγμή που θα συγκεντρώσει την παγκόσμια ενέργεια γύρω από την ισότητα των γενναιών. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο πρέσβης κύριος Εσκανιέρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Δικαιωμάτων της Γυναίκας, ε, ε, ε, κυρία Πρέσβη Πολιτικών Υποθέσεων της Γαλλίας και ε, κυρία Πρέσβη ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, αρμόδιας για τα γυναικεία ζητήματα. Είναι για μένα μεγάλη τιμή και χαρά να συμμετέχω με μεγάλο ενθουσιασμό σε αυτήν την εκδήλωση όπου θα εξετάσουμε πώς θα συγκεντρώσουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να προωθήσουμε μία, έναν από τους μεγάλες αγώνες της ανθρωπότητας, την ισότητα των φύλων. Ε, ε, σε αυτόν τον αγώνα η χώρα μου έχει παίξει ιστορικό ρόλο. Θα γνωρίζετε ότι στην πρώτη διάσκεψη που έγινε ε, το 1975 ε, για τα γυναικεία δικαιώματα συμβάλαμε σημαντικά όπως συμβάλαμε ε, και στην πλατφόρμα του Πεκίνου το 1995 και τώρα φιλοξενούμε την διάσκεψη αυτή τον Μάιο του 2020 και είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή αυτή τη στιγμή έχουμε τον πρόεδρό μας ε, που προωθεί μια ατζέντα προοδευτική, ε, γίνονται αλλαγές και η ισότητα των φύλων είναι στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Ε, Δηλαδή, προηγμένη νομοθεσία, ε, ε, ε, επίση με επικεφαλή στο Μαρίν Γκάσμαν το Ινστιτούτο για τις Γυναίκες δημιουργήθηκε και επίση είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε πραγματική ισότητα των φύλων τόσο στην κυβέρνηση όσο και στις διάφορες υψηλά ιστάμενες θέσεις. τα δύο σώματα ότι άνω και κάτω βουλή του Μεξικό προεδρεύονται αυτή τη στιγμή από γυναίκε. Αυτό είναι στοιχείο που μας γεμίζει με περηφάνεια. Και η εξωτερική μας πολιτική είναι πολύ φεμινιστική. Έχουμε βαθιά πεποίθηση, όπως τόνισε και ο καγκελάριος του Μεξικό, Μαρσέλ Γιγιάρ, στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον περασμένο Σεπτέμβριο. Έχουμε πολλά βέβαια ακόμα να κάνουμε σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Στο Μεξικό έχουμε, τερά... έχουμε τεράστιους στόχους σε αυτό το θέμα, τους οποίους ε, επιδιώκουμε με αποφασιστικότητα και σύμφωνα με την Ατζέντα 2030 και μέσω της διεθνούς συνεργασίας για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό και η ισότητα των φύλων είναι ένας οριζόντιος ε, άξονας που διέπει όλες μας τις πολιτικές. Όπως είχα την ευκαιρία να τονίσω και παλιότερα, η ιστορία του αγώνα για την ισότητα των φύλων μας δείχνει πως ε, οι στόχοι δεν είναι στατικοί. Πρέπει να ε, ε, γίνεται προσπάθεια διαρκής και μόνιμη, να είμαστε επίμονοι και υπομονετικοί γιατί για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους, γιατί ταυτόχρονα βλέπουμε και να γίνονται οπισθοδρομήσεις. Ε, πρέπει λοιπόν να είμαστε σταθεροί και πιστεύω πως ο ρόλος των κοινοβουλίων είναι πολύ σημαντικός σε αυτή την υπόθεση. Ως, ε, τα κοινοβούλια ως νομοθετικά όργανα, ως θεσμοί και ως επόπτες και ελεγκτές των τι συμβαίνει επί τόπου. Ε, γι' αυτό και πρέπει να δουλέψουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσουμε αυτή την ατζέντα, σίγουρα σε συνεργασία με την νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επίσης προσπάθησε να τηρήσει την ισότητα των φύλων, την ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την οποία αναπτύσσουμε έναν ε, πολυμερή διάλογο ε, το Μεξικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις κάναμε μια πρώτη συνεδρίαση τον Νοέμβριο για, για διάφορα πολυμερή ζητήματα με τη συμμετοχή της ε, <coughs> Μάρτα Ντελγάντο, υφυπουργού μας για τα διεθνή θέματα. Επίσης δουλεύουμε εντατικά για πολύ σημαντικά προγράμματα όπως το Spotlight που είναι ένα παράδειγμα για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα πολύ δύσκολα, σκληρά ε, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Ευρωκοινοβούλιο ε, ε, βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να εργαστούμε διμερώς αλλά και πολυμερώς και σε παγκόσμιο επίπεδο το Φόρουμ Ισότητας των Φίλων στο Μεξικό σε συνεργασία με την ε, ε, Ηνωμένα Έθνη Γυναίκες και στη συνέχεια με τη δεύτερη σύνοδο στο Παρίσι είναι ένα ανοιχτό φόρουμ για όλους όσους αγωνίζονται για την ισότητα των φίλων και σίγουρα για τους βουλευτές. Θέλουμε να έχουμε ατζέντα θετική, να δώσουμε θετική όθηση στις ε, παγκόσμιες <clears throat> διεθνείς προσπάθειες για την ανάπτυξη της βιώσιμης ε, ε, ανάπτυξης με πάντοτε με έξονα την ισότητα των ε, φύλων ώστε να υπάρξει μια θετική εξέλιξη μέχρι την επέτειο τη 25 ετών της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου. Και όπως σας είπα είναι πολύ σημαντικό για το Μεξικό το ότι φιλοξενούμε αυτή τη σύνοδο γιατί έτσι δείχνουμε πως είναι ένας παγκόσμιος αγώνας όπου μπορούν να συμμετέχουν όλες οι χώρες και όλες ιδιαίτερως οι αναπτυσσόμενες και οι αναδιόμενες χώρες μπορούν να συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο γιατί ε, Θέλουμε να κινητοποιήσουμε τους βασικούς ε, φορείς ε, που, για να συμμετέχουν στο Φόρουμ Ισότητας των Φύλων. Και ήδη έχει γίνει συζήτηση ανάμεσα στον πρόεδρο ε, Σασόλη του Ευρωκοινοβουλίου και την πρόεδρο της Διακοινοβουλευτικής Συνόδου που είναι αυτή τη στιγμή Μεξικανή ε, για να δούμε πώς μπορούν να συμμετέχουν έτσι ώστε τα κοινοβούλια να παίξουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του φόρουμ ε, για την ισότητα των φύλων που θα γίνει στο Μεξικό. Επίσης, ε, η ισότητα είναι θέμα κλειδί. Είναι κάτι επί το οποίο θέλουμε να δουλέψουμε εντατικά. Εκτιμούμε την ε, ηγεσία της Προέδρου της Επιτροπής σας με την οποία έχουμε έρθει σε επαφή διμερώς ήδη και ήθελα επίσης να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να επαναλάβω την πολύ θερμή μας πρόσκληση ε, ώστε η Επιτροπή σας, η Επιτροπή Δικαιωμάτων της γυναίκας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εκπροσωπηθεί στη χώρα μου. Θα μας βοηθήσετε πολύ και θα σας δεχτούμε με μεγάλη θέρμη. Να σας ε, ε, τονίσω επίσης ότι καλέσαμε τη Eurolat. Ε, επίσης έχουμε συζητήσει με τον Σύμπροεδρο Χαβιλόπες της, της με τη Eurolat, ώστε να αποτελέσουμε ως πρωταθλητές σε αυτό το θέμα. Και το ίδιο κάνουμε και με την μειχτή κοινοβουλευτική η Επιτροπή Μεξικό Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητάμε με τον πρόεδρο Μασιμιλιάνο Εσμερίγλιο και τα μέλη της Επιτροπής ε, και ε, ε, είδαμε μεγάλο ενθουσιασμό για τη συνεργασία και όπως σας είπα είμαστε σύμμαχοι στην <clears throat> προώθηση αυτού του θέματος διεθνώς. Σημαντική συμμετοχή βέβαια και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία επίσης ε, προσκαλούμε να συμμετέχει δραστήρια στο φόρουμ για την ισότητα των φύλων στο Μεξικό. Σας ζητούμε λοιπόν την υποστήριξή σας για να ε, προωθήσετε και εσείς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Επίτροπο Ισότητας και με την Επίτροπο ε, Διεθνών Σχέσεων και σίγουρα ε, και εσείς θα εξασφαλίσετε μαζί ε, μια μεγάλη εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το φόρουμ. Να επαναλάβω τέλος ότι σας περιμένουμε στο Μεξικό το φόρουμ ισότη... ισότητα των φίλων ε, στη χώρα μου θα είναι η πρώτη διάσκεψη που θα απηχήσει την πρώτη μάλλον διάσκεψη που έγινε το 1975 για τα δικαιώματα της γυναίκας στο Μεξικό. Ελπίζουμε πως θα είναι ένα μέγα βήμα μπροστά που θα προετοιμάσει τη Σύνοδο του Παρισιού, το δεύτερο φόρουμ που θα γίνει το φόρουμ και ελπίζουμε πως ο εορτασμός του Πεκίνου στο πλαίσιο του ΟΗΕ δεν θα είναι απλά μια επέτειος, αλλά θα είναι μια ουσιαστική προσπάθεια για παγκόσμια δέσμευση ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η ισότητα των φύλων θα μετατραπεί σε πραγματικότητα σήμερα, εδώ και τώρα μέσα στην Ατζέντα 2030. Αυτό είναι ο ιστορικός στόχος που έχουμε και η χώρα μου είναι απόλυτα προσιλωμένη και συμμετέχει και με την ε, πρεσβεία του Μεξικού εγώ και το προσωπικό μου θέλουμε προσωπικά να εκφράσω την προσωπική μου δέσμευση για αυτό ε, το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η πρέσβη της ε, Γαλλίας. Σας παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία mm. Γολά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, κύριε Πρέσβη. Πρώτα πρώτα σας ζητώ συγγνώμη από την Delphine, ε, εκ μέρους της Delphine O, της ε, πρέσβεως που θα έπρεπε σήμερα να σας ε, παρουσιάσει ε, το φόρουμ για μια ισότητα στο Παρίσι. Δεν μπόρεσε όμως λόγω της απεργίας που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Παρίσι να έρθει εδώ. Σας ζητάω εκ μέρους της συγνώμη. Και βεβαίως θα έρθει στις Βρυξέλλες με πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστούμε πολύ για την οργάνωση αυτής της συνεδρίασης. Ε, που ε, γιατί μπορώ και εγώ, όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές, να σας παρουσιάσω τι θα γίνει στο Παρίσι. Γνωρίζετε την δέσμευση της Γαλλίας υπέρ των δικαιωμάτων ε, των γυναικών, της ισότητας ανδρών και γυναικών, υπέρ της πολυμέρειας. Όλα αυτά βρίσκονται βεβαίως στο επίκεντρο, κυρίως λόγω της οπισθοχώρησης που διαπιστώνουμε όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών σε όλο τον κόσμο, παρόλη την πρόοδο που επιτέχθη μετά το Πεκίνο. Το φόρουμ λοιπόν αυτό ε, αφορά και το Μεξικό και τα Ηνωμένα Έθνη και το Παρίσι και για μας ε, είναι ο αγώνας που συνεχίζεται υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών για προώθηση της ατζέντα, για μεγαλύτερη συμμετοχή προκειμένου να επιτύχουμε συγκεκριμένους στόχους. Ε, από το Πεκίνο λοιπόν ε, και όλα τα επόμενα χρόνια θα συνεχιστεί η πρόοδος. Η Γαλλία δεσμεύεται ιδιαίτερα όσον αφορά αυτό, κυρίως όσον αφορά την προεδρία του G7 που ολοκληρώνεται και μετά λοιπόν την συνεδρίαση, μάλλον μετά το φόρουμ στο Μεξικό τον Μάιο, θα συνεχίσει το φόρουμ στο Παρίσι από τις 7 μέχρι τις 10 Ιουλίου 2020. Για μας λοιπόν θα είναι η ευκαιρία αλλά και για την UNIFAM αλλά και για το Μεξικό να συνεχίσουμε ε, αυτό που ονομάζουμε συνασπισμούς δράσης. Οι συνασπισμοί δράσης είναι μια συγκέντρωση ε, μεταξύ κρατών, ιδιωτικού τομέα, ε, πολιτών, προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι για να μπορέσουμε να ε, προοδεύσουμε, να εργαστούμε περαιτέρω ε, για το μέλλον. Έχουμε λοιπόν τον ιδιωτικό τομέα, τις κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και βεβαίως όπως είπαμε τα κράτη, διότι είναι κυρίως οι κυβερνήσεις οι οποίες στηρίζουν αυτούς τους συνασπισμούς. Τα ε, μήνυματα λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε να ακουστούν αλλά και οι συνασπισμοί αυτοί μπορούν λοιπόν να συνενώσουν τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα και να κάνουν να ακουστούν σημαντικά μηνύματα. Η διαδικασία λοιπόν για τη δημιουργία αυτών των συνασπισμών αυτή τη στιγμή ακόμα συνεχίζεται, δεν έχουν αποφασιστεί όλα, δεν μπορούμε λοιπόν να σας τα παρουσιάσουμε όλα ολοκληρωμένα. Ε, υπάρχουν ε, κάποιες θεματικές οι οποίες θα είναι εγκάρσεις ε, σε θέματα που θέλουν να προχωρήσουμε περισσότερο. Για παράδειγμα το κλίμα, την βία κατά των γυναικών, τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα και μετά την ε, υπουργική ε, διάσκεψη με το Μεξικό, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών που θα συμμετέχουν σε αυτούς τους συνασπισμούς δράσης, αλλά και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας και οι πολίτες, όλοι μαζί λοιπόν, ε, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα αυτών των συνασπισμών στα Ηνωμένα Έθνη τον Σεπτέμβριο. Έχουμε λοιπόν πολύ δρόμο μπροστά μας, πολύ δουλειά. Ε, πρώτον για να συγκροτήσουμε αυτούς τους συνασπισμούς, που όπως είπαμε είναι μια δουλειά που συνεχίζεται, θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες αλλά επίσης και για να κινητοποιήσουμε όλους τους παράγοντες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο να παίξει, τα θεσμικά όργανα, ξεκινώντας από την Επιτροπή, από το Ευρωκοινοβούλιο, όλοι συντελούν, αλλά Επίσης, ο καθένας μπορεί να μεταφέρει στη χώρα του το μήνυμα για την συμμετοχή του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα, για να τους κινητοποιήσουμε. Πρώτα λοιπόν στο Μεξικό και μετά στο Παρίσι, όλοι οι συμμετέχοντες, οι πιο σημαντικοί, θα δώσουν το παρόν. Ε, πάνω από 200.000 άτομα θα πάνε στο Μεξικό και 100.000 αναμένονται στο Παρίσι. Πολύ μεγάλη λοιπόν θα είναι η συμμετοχή. Η κινητοποίηση είναι για μας το πιο σημαντικό γύρω από αυτό το θέμα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι στο Παρίσι θα έχουμε σημαντικά αποτελέσματα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία και το 2025 να επιτύχουμε συγκεκριμένους στόχους, ε, ούτως ώστε να επιτύχουμε και τους στόχους της Ατζέντας 2030. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Μαρινάκη. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά από τρεις εξαίρετους ομιλητές, ε, Αναφέρθηκαν ήδη σημαντικά ε, στοιχεία, ο ρόλος μου επομένως είναι πιο εύκολος. Θα ήθελα να τονίσω όμως ιδιαίτερα την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς εμείς θα συμμετέχουμε σε ένα τόσο φιλόδοξο στόχο όπως το Φόρουμ Γενιά Ισότητα. Η κυριότερη πρόκληση για όλους μας έχει να κάνει με το 2020 διότι θα έχουμε πολλές σημαντικές επαιτίους που έχουν σχέση με θέματα ε, του θεματολογίου μας για τη χειραφέτηση των γυναικών, για την ισότητα των δύο φύλων και επίσης ε, για έναν απολογισμό όσον αφορά την ασφάλεια των ε, γυναικών. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μας να μπορέσουμε με ψυχραιμία να κάνουμε έναν απολογισμό για το τι επιτύχαμε όλα αυτά τα χρόνια. 25 χρόνια μετά το Πεκίνο, μετά την, ε, με το ψήφισμα για το 2025 και βεβαίως όσον αφορά το πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 2030. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν νομίζουμε ότι υπάρχει και κάτι επιπλέον. Υπάρχουν σημαντικές φιλοδοξίες για το Φόρουμ Γενιά Ισότητα για να μπορέσουμε, ε, να μπορέσουμε αυτόν τον απολογισμό να τον πάμε πιο πέρα και κυρίως για να έχουμε όλη μεγαλύτερη επίγνωση των ελλείψεων περισσότερο παρά των επιτυχιών μας. Βεβαίως και υπήρξε πρόοδος σε πολλά θέματα, Υπάρχουν ε, κάποια πράγματα που έχουν σήμερα προχωρήσει πολύ περισσότερο από ό,τι πριν από 25 χρόνια σίγουρα, αλλά οπωσδήποτε, όπως είπε και η αγαπητή φίλη κυρία Ντάγμαρ Σουμάχερ, θα πρέπει να αντιδράσουμε στην αντίδραση που συναντάμε. Η κατάσταση δεν είναι ιδανική ε, σήμερα, 40 χρόνια μετά, από ότι όταν ξεκίνησαν όλες αυτές οι προσπάθειες. Αλλά οπωσδήποτε δεν πρέπει να παραμένουμε ότι τα πράγματα στο μέλλον θα είναι πιο εύκολα για τα κορίτσια για τις γυναίκες. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι γενικότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά ιδιαίτερα τα δικαιώματα των γυναικών, στοχοποιούνται. Είναι πιο εύκολη στόχη μάλιστα μέσα σε κοινωνίες οι οποίες υποχωρούν σε από του είδους την αντίδραση. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μεγαλύτερη ηθική ευθύνη και να αγωνιστεί, να υπερασπιστεί αυτά τα δικαιώματα των γυναικών όχι μόνο μεταξύ των 28 κρατών μελών, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Είναι μια ευθύνη, λοιπόν, την οποία παίρνουμε ε, σοβαρά. Και γι' αυτό, λοιπόν, Στηρίζουμε ε, την πρωτοβουλία για μια ισότητα και θα συνεργαστούμε στενά τόσο με την Γαλλία όσο και με το Μεξικό και βεβαίως με όλους τους συμμετέχοντες, με το UN Women, με τους, τις συναδέλφους μας, τους συναδέλφους μας εκεί, για να έχουμε μεγάλη επιτυχία, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλά που θα πρέπει να προωθηθούν, να έρθουν στο προσκήνιο και ότι η πρωτοβουλία Γενιά Ισότητα πραγματικά αξίζει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ε, θα ε, προσδιορίσει και τη νέα ανανεωμένη μας προσέγγιση, η οποία αποτυπώνεται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόεδρο Ursula von der Leyen, αλλά και με τις ε, πέντε επιπλέον επιτρόπους και αντιπροέδρους της Επιτροπής ε, που συμπληρώνουν ε, που, την Επιτροπή και που αναλαμβάνουν καθήκοντα για την χειραφέτηση και τα δικαιώματα των γυναικών σε όλους τους τομείς. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική δέσμευση την οποία θέτουμε στην υπηρεσία της πρωτοβουλίας για μια ισότητα. Σκοπεύουμε λοιπόν να ε, στηρίξουμε τους συνασπισμούς δράσης και έχουμε ήδη ένα πλαίσιο ε, μέσω, ε, δράσης μέσω της πρωτοβουλίας Spotlight, όπως είπε και ο πρέσβης Εσκανέρο. Είναι μια παγκόσμια προσπάθεια για να καταργηθεί κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και σε συγκεκριμένες περιφέρειες και μέρη του κόσμου, όπου προσπαθούμε σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών και όλους τους σημαντικούς ε, εταίρους, να επιταχύνουμε ε, την πρόοδο, η οποία έχει ήδη καθυστερήσει, ε, για την κατάργηση της βίας κατά των γυναικών που μαστίζει ε, τις γυναίκες σε πολλές κοινωνίες. Η βία κατά των γυναικών λοιπόν είναι ένας τομέας όπου οπωσδήποτε ο συνασπισμός, ε, οι συνασπισμοί δράσης θα κάνουν τη διαφορά, θα δεσμευτούμε οπωσδήποτε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου θα δεσμευτούμε ισχυρά. Αναμένουμε λοιπόν ε, το σχετικό έγγραφο, το οποίο θα προκύψει, ελπίζουμε να το έχουμε στο δυνατό γρηγορότερα, προκειμένου να το εξετάσουμε προσεκτικότερα και να ε, δεσμευτούμε πιο συγκεκριμένα. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό επίσης να τονίσουμε ότι θεωρούμε πολύ σημαντική, ε, σημαντικό σε αυτή την πρωτοβουλία να αποφευθούν οι αλληλεπικαλύψεις να ε, επιδιώξουμε μια συμπληρωματικότητα δράσεων ε, και κυρίως ε, όλα τα, όλα τα θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχουν ενεργά και να στηρίξουν την πρωτοβουλία με κάθε δυνατό τρόπο. Και τέλος, το 2020 από πλευράς μας εμείς ετοιμαζόμαστε στην νέα επιτροπή. Είμαστε όλοι ενθουσιώδες με αυτό για να έχουμε μια νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και νομίζω ότι θα, στο πρώτο εξάμεινο του 2020 θα την έχουμε κιόλα. Η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν και η Έλενα Ντάλι, νέα επίτροπος για την ισότητα των φύλων, έχουν δεσμευτεί και βεβαίως θα, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε την πρωτοβουλία να επιτύχουμε χρηματοδότηση εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να μπορέσουμε έτσι να ε, διευρύνουμε το πεδίο, να εμπλέξουμε περισσότερες χώρες και να καλύψουμε περισσότερους τομείς που έχουν σχέση με τη βία κατά των γυναικών που θέλουμε να καταργήσουμε. Και έχουμε ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις και προσβλέπουμε επίσης ε, και στην συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο την πολύ σημαντική επικοδομητική του συμβολή για το επόμενο σχέδιο δράσης για τα φύλλα. Είναι ένα σχέδιο δράσης που θα διαδεχθεί το σημερινό σχέδιο δράσης, θα διευρύνει το πεδίο του και θα προσθέσει νέους στόχους. Για όλα αυτά λοιπόν προσβλέπουμε σε εσά στη στήριξή σας σε όλους σας να στηριχθείτε, να μας στηρίξετε μάλλον, να δεσμευτείτε για να καλυτερέσουμε τη ζωή ε, εκατομμυρίων γυναικών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές μας. Και τώρα η κυρία Χενρίτα Γκάγκερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και λυπούμε που καθυστέρησα. Είχα κολλήσει σε ένα σανσέρ στο κτίριό μας. Πολύ θα ήθελα να βρισκόμουν εδώ και για το σημείο ICPD, για τη Σύνοδο, για τον πληθυσμό, όπου είχαμε μια πολύ ισχυρή παρουσία ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να επαναληφθεί και στο μέλλον, για αυτά που προσπαθούμε να επιτύχουμε ε, έως το 2020. Οι προηγούμενοι ομιλητές ήδη επεσήμεναν τα περισσότερα από τα σημεία που ήθελα και εγώ να θίξω, ιδίω η Μάρα, Οπότε θέλω να πω ότι η πλήρης αφοσίωση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ισότητα των φύλων. Το είδατε με τις δηλώσεις της Προέδρου Φοντερ Λάιν, της κυρίας Γιούπι Λάινεν. Η νέα μας Επίτροπος ε, είναι ταγμένη στο σκοπό τη ισότητας των φύλων. Και θα προσπαθήσει να προωθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα θέματα αυτά κατά τη διάρκεια της θητείας της. Με χειροπιαστή συνεργασία αλλά και με την δική της την παρουσία και το πολιτικό της βάρος. Και όπως είπα, ε, εσωτερικώ κάνουμε μια αξιολόγηση για την ισότητα των φύλων. Αυτό θα ε, συμπληρωθεί από τον GAP 3, οπότε εσωτερικώ στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουμε μια καλή βάση. Είναι ένα καλό εφαλτήριο θα πρέπει λοιπόν να το ε, δούμε αυτό σε μια πρώτη φάση με προσοχή. Είναι ένα πρώτο σημείο σύγκλησης με το ε, Φόρουμ για την Ισότητα των Φύλων. Ε, περιμένουμε ακόμα που θα χρειαστεί συνεννόηση, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η προστιθέμενη αξία, που εμείς ως θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να έχουμε προστιθέμενη αξία. Και θέλουμε να συμμετέχουν όλοι, άντρες και γυναίκες. Δεν μας παίρνει δεν μπορούμε πλέον να μην αναζητούμε οποιοδήποτε συνασπισμό για το θέμα αυτό και να δεχτούμε πιστοδρομήσεις ή υπαναχωρήσεις. Μόλις λοιπόν έχετε κι εσείς ξεκαθαρίσει τις ιδέες σας, θα πρέπει να προσθέσουμε τη φωνή μας στην, ε, στο συνασπισμό τη συμμαχία για τη δράση, ίσως για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών, θα δούμε που μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερη προστιθέμενη αξία και απλώς να πω το εξής. Για να πετύχουμε χρειαζόμαστε και την κοινωνία των πολιτών στο πλευρό μας. Όπως είπε και ο πρέσβης από το Μεξικό, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αλλαγή του, των προτύπων που ισχύουν στην κοινωνία, με τις νόρμες. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει στην κοινωνία, γι' αυτό χρειάζεται μια συμμαχία ως το δυνατόν ευρύτερη, ε, όσο το δυνατόν περισσότερο. Και όπως είπε και εκπρόσωπος από την Γαλλία χρειάζεται και ο ιδιωτικός τομέας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν ε, τώρα, το 2020 δηλαδή, να προσπαθήσουμε να, να έχουμε μια ισχυρή, μια δυνατή φωνή ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όλα τα κράτη-μέλη. Μόνον έτσι θα επιτύχουμε το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε. Γι' αυτό παρακαλώ στηρίξτε πλήρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία τα λόγια σα. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγο στου ε, βουλευτέ. Η Φράνση, η Χρυσούλα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ όλους ε, για τις ομιλίες σας και τις παρουσιάσεις σήμερα το πρωί. Ήθελα να πω ότι είναι ενθαρρυντικό να ακούμε τι επίπεδο φτάνει η αφοσίωσή μα και τι ειδικέ γνώσει έχει το καθένα από εσά. Ε, είναι πολύ καθησυχαστικό να τα ακούμε αυτά σήμερα το πρωί και ευχαριστούμε για τι συνεισφορέ σα κάθε μια από τι οργαν... Ε, από τις οργανώσεις σας, από τις ενώσεις σας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το Μεξικό ε, και επειδή έχω εργαστεί κατά θέματα αυτά εδώ και 20 χρόνια, πραγματικά με χαροποιεί. να πω ε, στο βέβαια από το Μεξικό, ότι πήγε μια Ιρλανδή ε, σε μια από τις διασκέψεις στο Μεξικό τη δεκαετία του 70 και ε, αν συγκρίνω τώρα τι φοβερή πρόοδος έχει γίνει, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Δηλαδή, θυμάμαι τι μα είχε πει γυρνώντα τότε στην Ιρλανδία από την πρώτη διάσκεψη και πραγματικά είναι πολλά τα βήματα πρόοδου. Ε, και αυτό ελπίζω να γίνεται σε κάθε χώρα. Εγώ τα θυμάμαι από τότε που τα είχα πρώτα ακούσει. Κάποιε γενικέ παρατηρήσει τώρα. Ε, πολλά υπόθηκαν, αλλά μερικά βασικά σημεία για το τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη φάση. Εάν σκεφτούμε τα θέματα ισότητας των φίλων των γυναικών, κάποτε ο κόσμος πίστευε ότι υπάρχει ουσιαστικά ένας ε, σκοπός που πρέπει να εκπληρωθεί για το θέμα αυτό. Δηλαδή ότι πρέπει να πετύχουμε ένα τόσο ποσοστό δικαιωμάτων και μόλις γίνει αυτό θα πάψει η συζήτηση. Αυτό δεν ισχύει πια με την παγκόσμια διάσκεψη. Βλέπουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν διαρκώς, υπάρχουν νέες μορφές, νέες ανάγκες, ε, νέες απαιτήσει. Και αυτό είναι σημαντικό το φόρουμ για την ισότητα των γενεών από μόνο του, αλλά χρειάζεται και μια ανανεωμένη, μια καινούργια προσέγγιση. Πρέπει μερικά πράγματα να τα ξανασκεφτούμε, αλλά υπάρχουν και νέα θέματα που έχουν ε, ανακύψει τώρα, έχουν ε, τώρα να δυθεί. Για την ευρύτατη συμμαχία, όντω έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Χρειάζεται μια, ευρύτερη, μια στο δυνατόν ευρύτερη συμμαχία, να βεβαιωθούμε ότι συμμετέχουν νέοι άνδρες και γυναίκες και μετά γι' αυτό είναι σημαντική η διάσκεψη αυτή, όλες αυτές οι διασκέψεις και γι' αυτό πρέπει να έχουμε κυρίως συνομιλίες. Τα είπαμε προηγουμένως για το τι έκαναν οι ΙΠΑ στο Νερόμπι για, την, για τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο και ένα επίπεδο πολιτική ηγεσία να αναλάβουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Το έχουμε δει αυτό μέσα από τι δεκαετίε. Η πολιτική ε, ασκεί μεγάλη επίδραση και αλλάζει τα πράγματα. Είναι σημαντικό το πώ οι γυναίκε ε, ε, μπορούν να προβληθούν μέσω των βασικών πολιτικών δεσμεύσεων στο ε, ανώτατο δυνατό επίπεδο. Μέσω αυτή τη διάσκεψη και όλων των ανάλογων. Ε, δεν πρέπει να τα υποτιμούμε αυτά. Ακούσατε να λένε οι Κλίντον στο Πεκίνο ότι γίνεται με τα γυναικεία δικαιώματα. Είναι δικαιώματα δημοκρατικά, θεμελιώδη δικαιώματα. Και εδώ δεν μιλάει εκ μέρου όλων, αλλά θέλω να φτάσω και στο εξή. Ε, είναι σημαντικό να τα προβάλλουμε και σε εθνικό επίπεδο όσα γίνονται. Διότι δεν νομίζω ότι πολλοί γνωρίζουν, δεν θέλω να προσβάλλω κανένα λέγοντα το αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι πολλοί γνωρίζουν ε, στο επίπεδο των απλών ανθρώπων, των απλών πολιτών, τι γίνεται με την ισότητα των φίλων, των γενεών και τι γίνεται με τις διασκέψεις. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το καθεξής να ε, περάσουν ένα ισχυρό μήνυμα για, αυτά τα, για αυτές τις διασκέψεις, για τη διάσκεψη συγκεκριμένα αυτή και τις ανάλογες. Δηλαδή πρέπει να πετύχουμε χρηματοδότηση το Πεκίνο. Ε, είχε μεγάλη διεθνή αναγνώριση. Είναι σημαντικό ε, να δούμε τι αλλαγέ μπορέσαμε να πετύχουμε χάρη σε, τέτοιες σε αυτή την προβολή και κάτι ανάλογο να γίνει σε όλες αυτές τις διασκέψεις. Νομίζω ότι χρειάζεται και μια νέα παρουσίαση του θέματος για να βεβαιωθούμε ότι ο κόσμος συνεχίζει να ενδιαφέρεται, να παθιάζεται για τα θέματα αυτά και να δίνει σημασία στα ζητήματα και την ανάγκη να κάνουμε κάτι για αυτά. Χρειάζεται λοιπόν αφοσίωση και δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχετε πολύ καλό κατάλογο προτεραιοτήτων, πολύ καλή ατζέντα, έχετε τις απαραίτητες ε, γνώσεις και πιστεύω ότι θα έχουμε και τα στατιστικά στοιχεία. Πρέπει να υπάρξει διεθνής ε, επικέντρωση στα γυναικεία δικαιώματα. Η διάσκεψη στο Ναϊρόμπι ήταν ε, πραγματικά βάσει των στοιχείων που είδαμε κάτι που μα αναστάτωσε. Δηλαδή σε τόσα μέρη του κόσμου να υπάρχει τέτοια υποβάθμιση των γυναικείων δικαιωμάτων. Πρέπει βεβαίω να αναγνωρίσουμε και την πρόοδο που έχει γίνει. Θα ήταν ε, ανεύθυνο από μέρο μα να μην το κάνουμε. Αλλά υπάρχει και πολιτική οπισθοδρόμηση. Και ταυτόχρονα για να συνεχίσουμε να τους έχουμε στο πλευρό μας, όσους δεν είναι οι πρώτοι ε, που συμμετέχουν, ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε και την πρόοδο. Χρυσούλα. Ευχαριστώ, Ευλίν. Ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές μας σήμερα το πρωί. Πραγματικά χαίρομαι πολύ ως νέο μέλος του Κοινοβουλίου, προερχόμενο από τη Γαλλία, να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Βλέπουμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο Μόλις επιστρέψαμε από τον Ναϊρόμπι, βλέπουμε ότι υπήρχε ένα, μια συνολική δέσμευση όλων, ασχέτως πολιτικής ομάδας, να προωθήσουν τον ίδιο σκοπό και εδώ πραγματικά όλοι ενδιαφερόμαστε να ε, αναβαθμίσουμε το θέμα των γυναικείων δικαιωμάτων. Η Επιτροπή Γυναικών τα έχει, συνεχί... τα έχει συζητήσει διαμακρών, τα έχουμε συζητήσει και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω όμως τώρα να χαιρετήσω τις δεσμεύσεις της νέας επιτρόπου. Της νέας επιτρόπου για τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις, για την ανάπτυξη, γιατί η κυρία Γιούτα Ορπιλάινεν ε, κατά τη διάρκεια των ακροάσεων της ε, δεσμεύτηκε ώστε το GAP 3 να προχωρήσει. Αυτό καλό είναι να υπογραμμιστεί εκείνη θα αναλάβει να ε, υλοποιήσει τα προγράμματα αυτά και η Επιτροπή της Ανάπτυξης θα τα ε, φέρει στο φως της εξέτασής της και θα πρέπει η Επίτροπη Νταλή και Ουρπιλάινεν να εργαστούν από κοινού ώστε να ε, φέρουν στο προσκήνιο και σε πρώτη θέση τις ευρωπαϊκές αξίες, όχι μόνο εδώ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Το είδαμε, το Human Peace and Security. Ε, το θέμα που ανέφερε η κυρία Μαρινάκη. Είναι ακόμη μια δοκιμασία που θα πρέπει να δείξει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση καταφέρνει να προωθήσει τις αξίες της. Για το Μεξικό, τη διάσκεψη αυτή και τα όσα έγιναν στο Παρίσι, αυτή η συνέχεια, αυτή η εξακολούθηση τη ε, εξέταση των θεμάτων από μια διάσκεψη στην άλλη είναι σημαντικό γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια η κοινωνία των πολιτών, νέοι, άντρε και γυναίκε, δραστηριοποιούνται πολύ για να προωθήσουν την ισότητα. Τώρα λοιπόν πρέπει εμείς από τη δική μας τη θέση και οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων πραγματικά να δεσμευτούν και να αναλάβουν δράση. Και εάν μου επιτρέπετε, όπως και ο πρόεδρός μου, ο κύριος Μακρόν, πρέπει να το κάνουμε αυτό ένα θέμα εθνικό. Πρέπει κάποια στιγμή παντού στον κόσμο ε, να μην είναι μεμονωμένη η εξέταση των θεμάτων αυτών. Πρέπει να συμμετέχει ολόκληρη κοινωνία, ξεκινώντας από το εκπαιδευτικό σύστημα, από τα σχολεία, για να περάσουμε στην ε, εκπαίδευση των γενεών και κάποια στιγμή στο μέλλον οι μελλοντικέ γενναίε να θεωρούν κάτι το αυτονόητο την ισότητα ανδρών και γυναικών. Και να ολοκληρώσω λέγοντα ότι το Ευρωκοινοβούλιο και οι επιτροπέ ε, δικαιωμάτων των γυναικών και ανάπτυξη θέλουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Θέλουμε να οργανώσουμε εκδηλώσει στο περιθώριο και πραγματικά χαιρόμαστε πολύ που μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη ε, διάσκεψη για τα δικαιώματα των γυναικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ η κυρία Jones και μετά η Μαρία Μανουέλ. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ευχαριστήθηκα πολύ τις ομιλίες σας και τις συνεισφορές σας και πραγματικά πήρα κουράγιο. Γιατί έχουμε τέτοιες δεσμεύσεις ε, υψηλό πολιτικό επίπεδο ε, στο πρόγραμμα. Ε, τώρα, ένα σχόλιο, μια ερώτηση για την Dagmar για την επόμενη χρονιά, το CSW. Ακούσαμε ότι είναι μια σημαντική χρονιά από πολιτική σκοπιά. Και όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν ταυτόχρονα, όλες αυτές οι διασκέψεις. Πριν από πέντε χρόνια, επίσης είχαμε την πολιτική δήλωση στην ε, αντίστοιχη διάσκεψη. Καλό είναι να έχουμε, όπως είπαμε, ευρύτατη συμμαχία με συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, αλλά βλέπουμε να συρρυκνώνεται η, συμμετοχή το, ποσο, το ποσοστό συμμετοχή με την αποχώρηση των ΗΠΑ με όσα έγιναν στο CSW, ότι το χρήμα στερεύει και αυτό που διατίθεται στην κοινωνία των πολιτών. Το λέω λοιπόν, κάντε ό,τι μπορείτε. Ε, ε βλέπουμε ότι ό,τι ξοδεύει κανείς φέρνει περισσότερους ακτιβιστές. Πάντως για τη συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών. Πώ μπορούμε να το βάλουμε αυτό και στο ε, σχέδιο τη πολιτική δήλωσης γιατί είναι τόσο σημαντικό πολιτικό έτο από πολλέ διαφορετικέ απόψει. Ε, είναι σημαντικό να έχουμε μεγάλη συμμετοχή βέβαια, αλλά θέλουμε να τους φέρουμε αν γίνεται ως εκεί. Είναι πολύ ε, ακριβό, πολύ, κοστίζει πολύ αυτές οι οργανώσεις να καταφέρουν να έρθουν ως εκεί και να συμμετέχουν. Και το θέμα είναι να μην έχουμε πάντοτε του ίδιου συμμετέχοντε, του ίδιου φορεί κάθε χρόνο από τη μια διάσκεψη στην άλλη, γιατί ακούγονται ίδιε φωνέ γύρω από το τραπέζι και οι ίδιε φωνέ. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε μια πολυφωνική ε, προσέγγιση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για τις συνεισφορές. Θα τα πω πορτογαλικά. Ευχαριστούμε, χάρη στους Γερμανείς μάλλον. Είναι σημαντικές οι ε, κοινέ μας προσπάθειες. Πρέπει να αποφύγουμε τις επαναλήψεις, διότι τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι σοβαρότατα και είναι κοινά για όλους μας, σε πολλούς ε, από τους τομείς της δραστηριότητάς μας και σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Ακούσαμε πολλά προβλήματα να θίγονται εδώ, προβλήματα που θεωρούσαμε ότι είχαν ήδη επιληθεί από τον προηγούμενο αιώνα, όπως της οικογενειακής βίας ή του ακροτηριασμού των γενικών, γενετικών οργάνων. Αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως. Δυστυχώς όμως παραμένουν προβλήματα για τα οποία δεν έχουμε κινητοποιήσει ακόμα αρκετά τις δυνατότητες που θα έπρεπε. Γι' αυτό και η συζήτηση για τον αερόμπι που έγινε μόλι προηγουμένω. Δυστυχώ επίση για... είναι προβλήματα για τα οποία δεν έχουμε εξεύρει την κατάλληλη λύση. Και πρέπει να το πούμε αυτό με κάθε ταπεινοφροσύνη. Δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε αντιστρέψει την ε, τάση. Ε, σα ίσα βρισκόμαστε απλώς σε πορεία αντιστροφής αυτής της τάσης. Θα χρειαστεί όμως καιρός και αυτό πρέπει να πούμε. Πρέπει να εργαστούμε ε, μαζί, συλλογικά, για να αναζητήσουμε λύσεις. Η λύση θα είναι περίπλοκη, πολυδιάστατη και θα απαιτήσει την κινητοποίηση πολλών διαφορετικών δυνάμεων. Και θα πρέπει κάποιες φορές να έχουμε καλύτερη αντίληψη των προβλημάτων. Γι' αυτό θα πρέπει να συζητάμε τα δεδομένα και τα στοιχεία. Πολλές φορές δεν έχουμε καν τις ε, απαραίτητε πληροφορίες για να κατανοήσουμε τις διαστάσεις ενός προβλήματος. Και αν δεν το αντιληφθούμε σωστά, αν δεν το κατανοήσουμε, δεν θα βρούμε και τη σωστή λύση. Ταυτόχρονα όμως, και νομίζω γι' αυτό το φόρουμ πρέπει να δώσει μια όθηση στην εξέταση των προβλημάτων του νέου αιώνα, πρέπει να δούμε και τις νέες ισορροπίε, ε, τα νέα προβλήματα που αναδύονται. Εάν δεν τα προλάβουμε τώρα, θα ε, γίνουν πολύ σοβαρότερα, θα οξυνθούν στο μέλλον. Όπω αυτό αυτό που ε, είδαμε πρόσφατα και το βλέπει και η συνάδελφος Λίνα Ταλβές. Δηλαδή την άνεση εκπροσώπηση των γυναικών σε επαγγελματικούς κλάδους, τα μελλοντικά επαγγέλματα. Αυτά που σχετίζονται κυρίως με τις νέες τεχνολογίες, με την πληροφορική. Και πρέπει εδώ να υπάρξει πληροφόρηση και εκπαίδευση. Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση πρέπει να είναι θέμα που θα συζητηθεί στο φόρουμ ε, και πραγματικά ευχαριστώ πολύ τον ε, πρέσβη για τον ενθουσιασμό του, για το πάθος του. Έχουμε και την ερχόμενη εβδομάδα ένα φόρουμ που θα ασχοληθεί με τα θέματα αυτά στο επίπεδο του Eurolat. Ευχαριστούμε και την Πρέσβη από τη Γαλλία και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω αν εργαστούμε από κοινού, ίσως κάτι να καταφέρουμε να κάνουμε και θα ε, ε, είμαστε και ευτυχέστεροι ω μέλη αυτή τη Επιτροπή, πάνω από αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει απολύτω. Ευχαριστούμε. Λίνα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Ε, ήταν για λόγους ιατρικούς. Δεν άκουσα όλη τη συζήτηση. Απλώς ε, για την εκπρόσωπο της Επιτροπής. Μόνο εκείνη πρόλαβα να ακούσω και ήθελα να το σχολιάσω. για τις δεσμεύσεις της νέας Επιτροπής ε, ως προς την ισότητα των φύλων. Είπατε κάτι που είναι σημαντικό και συχνά το ξεχνάμε. Λέτε ότι θα εργαστείτε για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. Ε, ως τώρα, τι έχουμε δει στην οικονομική σφαίρα, στις πολιτικές, τις δημοσιονομικές και οικονομικές. Περισσότερο πολιτικές απασχολησιμότητας παρά ισότητας. Είναι διαφορετικά αυτά. Και είναι σημαντικό γιατί γυναίκες και άνδρες ε, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και μετά μπορούν να κάνουν μια σταδιοδρομία, αλλά με πολύ διαφορετικούς τρόπους, άνισους, για να το πω έτσι. Και εάν κοιτάμε μόνο την απασχολησιμότητα, δεν θα γίνει αλλαγή. Πρέπει να μπει και η παράμετρος της ισότητας στο οικονομικό και στο μακροοικονομικό επίπεδο και στις πολιτικές μας. Αυτό δεν συμβαίνει καθόλου. Δεν υπάρχει κανένας προσανατολισμός προς την ισότητα των φύλων. Ναι. Τίποτε το σχετικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο πολιτικές λιτότητας επιβάλλονται. και μάλιστα έχουν λειτουργήσει κατά των γυναικών στην πραγματικότητα και εντελώ ξεκάθαρα. Φυσικά έχουν πλήξει πολύ κόσμο, αλλά όλο ιδιαίτερο τι γυναίκε. Οπότε πρέπει να υπάρξει μια ευθυγράμμιση της διάστασης των φύλων στην καρδιά των οικονομικών μας πολιτικών. Όχι μόνο για την Ευρώπη και για άλλες περιοχές του κόσμου. Διότι οι πολιτικές λιτότητας εφαρμόζονται και αλλού. Και εδώ ίσως είμαστε και σε ευνοϊκότερη θέση για να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Σκεφτόμενοι, συλλογιζόμενοι την αυστηρός οικονομική πολιτική. Μην μείνουμε στις κοινωνικές πολιτικές, στις πολιτικές ισότητας ή τις πολιτικές απασχολησιμότητας ε, ξεχωριστά. Εάν θέλουμε οικονομική χειραφέτηση πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πιερέτ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους ε, ομιλητές που έκαναν ε, σπουδαίες δηλώσεις και διαπιστώνουμε μεγάλο ενθουσιασμό και κυρίως δέσμευση και ευχαριστώ όλους ιδιαίτερος τον πρέσβη του Μεξικού και της Γαλλίας. Όμως ακούμε επίσης ε, εδώ τη φωνή των γυναικών που δεν τις ακούμε συχνά και σκέφτομαι όλες τις μετανάστριες που βρίσκονται στις ε, ευρωπαϊκές χώρες και θα πρέπει να ε, πολύ συχνά δεν αποτελούν τμήμα αυτής της μεγάλης διεθνούς επαφής. Αυτή τη στιγμή έχουμε την Επίτροπο για την εταιρικότητα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε και αυτή την εταιρικότητα για τις χώρες τις οποίες για τις γυναίκες τις οποίες ξεχνάμε και που επίσης αγωνίζονται για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και πολύ συχνά έχουν προβλήματα με κουλτούρες ε, διαφορετικές. Ε, τα προβλήματα δηλαδή είναι εγγενή στην ε, κουλτούρα προέλευσής τους. Θα πρέπει λοιπόν να καλλιεργήσουμε αυτό το πρόσωπο της επικοινομορφίας και ε, η κυρία Γκάλη μας το συζήτησε πολύ ότι δηλαδή θέλει ε, αυτή η πολυμορφία να ισχύσει ανάμεσα στις οργανώσεις και... θα κοιτάξουμε να ε, συνδυάσουμε και άλλες φωνές που ακούγονται όπως είπε και η συνάδελφος για να υπάρχει πολυφωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Πρωτού δώσω το λόγο στους ομιλητές μας για να απαντήσουν, μία ερώτηση απευθεία στην κυρία Σουμάχερ. Μιλήσατε για satellite sessions, για τις δορυφορικές ε, συνόδους. Πώς θα οργανωθεί αυτό, μπορείτε να μας πείτε περισσότερα. Και μετά για την ερώτηση που θέσατε πολλέ από εσέ, το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Το Μεξικό δεν είναι και δίπλα. Το Παρίσι είναι άλλο, αλλά για κάποιου και αυτό είναι μακριά. Πώ θα μπορούσαν να συμμετέχουν με κυβερνητικέ οργανώσει που δεν έχουν ε, αρκετά κονδύλια. Να ξεκινήσουμε με την ίδια σειρά όπω ε, τοποθετηθήκατε. So much. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια πολύ ε, πλούσια συζήτηση. Μακάρι να είχαμε ώρες και ώρες για να εξαντλήσουμε το θέμα. Αλλά θα ξεκινήσω απαντώντας στις ερωτήσεις που μου έγιναν απευθείας. Και μετά ίσως θα εκφράσω και κάποιες σχέσεις, ε, σκέψεις. Όσον αφορά λοιπόν την ερώτηση της Jackie Jones, Έχουμε λοιπόν το Προεδρείο του CSW που έχει κάνει μια συζήτηση στις 11 Δεκεμβρίου ίσως θα συνέλθει για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω με πολιτική δήλωση. Θα επανέλθω λοιπόν, αλλά θα ήθελα απλώς να σας πω ότι ήδη το θέμα συζήτηται. Ακούμε λοιπόν τη φωνή της κοινωνίας των πολιτών. Βεβαίως ε, οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών σε όλο τον ε, κόσμο ενδιαφέρονται. Υπάρχει το site μας ε, όπου μπορούν όλοι να επισκεφθούν. Επίσης, θέλουμε να παροτρύνουμε όλες τις αντιπροσωπείες των χωρών να συμπεριλάβουν στις αναχώρα αντιπροσωπείες τους μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Το είπατε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω λοιπόν ότι θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών ε, φέτος από τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, όσον αφορά το Φόρουμ για μια ισότητα, υπάρχει ένας μηχανισμός ε, για να συμπεριλάβουμε την κοινωνία των πολιτών. Αυτό απαντά και στην ε, ερώτηση της ε, Εύελιν. Δηλαδή, ποια είναι η δομή διακυβέρνησης του φόρουμ, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει μια κύρια ομάδα με τη Γαλλία, το Μεξικό, το UN Women και με εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών. Ε, είναι λοιπόν ένας χώρος που μπορεί να ακουστεί έντονα η φωνή της κοινωνίας των πολιτών. Μετά υπάρχει μια ομάδα συμβουλευτική της κοινωνίας των πολιτών με μέλη της κοινωνίας των πολιτών και επίσης υπάρχει και ε, μια διευθύνουσα επιτροπή ε, με συμμετοχή πολλών διαφορετικών παραγόντων. Επομένως υπάρχει έντονη συμμετοχή από όλο τον κόσμο της κοινωνίας των πολιτών όπως πολύ σωστά ζητήσατε. Τώρα όσον ε, αφορά αυτές τις συνδέσεις μέσω δορυφόρου, αυτό που εμείς θέλουμε είναι ε, να συμμετέχουν λοιπόν οι χώρες με αυτόν τον τρόπο στους συνασπισμούς δράσεων και να υπάρξει εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών διαγενειακή. Το 25% των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών είναι νέοι, από οργανώσεις από όλο τον κόσμο. Και βεβαίως εδώ σημαντική είναι και η τεχνολογική πτυχή. Θα γίνει λοιπόν μια συζήτηση μεταξύ πολλών διαφορετικών χωρών. Ομάδες χωρών θα συμμετέχουν σε αυτό το φόρουμ ε, και έτσι η συζήτηση αυτή θα γίνει ακόμα πιο διεθνής. Και βεβαίω για όλε αυτές τις ε, δορυφορικές συνδέσει διασκέψεις μέσω δορυφόρου και στο Μεξικό και στο Παρίσι θα υπάρχουν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων, ε, πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα είναι λοιπόν η συμμετοχή πραγματικά πολυπλευρική. Θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ, να συγχαρώ την Επιτροπή σας, ΦΑΜ, διότι οργανώσατε αυτό την συζήτηση αυτού του θέματος μετά τη συζήτηση για το ICPD. Νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να πάμε πιο πέρα. Νομίζω ότι και οι δύο εκδηλώσεις συνδέονται μεταξύ τους και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ενωριέτε Γκάιγκερ που ήταν μια πολύ δραστήρια παρουσία στο Ναϊρόμπι. Επίσης, κάτι που παρέλειψα να σας πω προηγουμένως, μετά το φόρουμ στο Παρίσι ε, θα υπάρξει και μια γενική, θα γίνει και μια γενική συνέλευση που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το φόρουμ Πεκίνο συν 25 τον ε, Σεπτέμβριο. Παρακαλώ να το σημειώσετε ήδη από τώρα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση για την στήριξή της ε, στις, στους συνασπισμούς δράσης. Για μας ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε στήριξη για αυτές τις δράσεις και ελπίζω να κατορθώσουμε έτσι να θέσουμε ένα τέρμα στη βία κατά των γυναικών. Και βεβαίως πολύ σημαντική είναι και η πρωτοβουλία Spotlight όπως είπε και η Ανριέτε Γκάιγκερ, είναι μια άριστη ευκαιρία να διευρύνουμε το πεδίο Spotlight, να, η πρωτοβουλία αυτή να πάει και σε άλλες χώρες, να εμπλέξουμε και άλλες ε, περιοχές του κόσμου και να έχουμε έτσι ένα πιο δυναμικό κίνημα. Θα ήθελα επίσης ε, εδώ, στο πλαίσιο της συζήτησης ε, ε, για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών, να ευχαριστήσω τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στις 25 Νοεμβρίου έδωσαν ένα πολύ δυναμικό παρόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε δυναμικό παρόν, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Συμβούλιο, πολλές αντιπροσωπείες σε όλο τον κόσμο δραστηριοποιήθηκαν στις διάφορες πρωτοβουλίες για την βία κατά των γυναικών, για την καταπολέμησή της και θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι επίσης όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κομισιόν και την ατζέντα για την ισότητα των φύλων. Προσβλέπουμε λοιπόν σε στενή συνεργασία μαζί της. Και θα ήθελα επίση να προσθέσω κάτι για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι βεβαίως μια άριστη ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε θέματα ισότητας των φύλων, να συμπεριλάβουμε τη διάσταση του φύλου στον προϋπολογισμό και βεβαίως υπάρχει δέσμευση της Κομισιόν για περαιτέρω πρόθεση της ατζέντα. Θα ήθελα εν συντομία να ε, επενέσω την, τον στο χαρακτηρισμό του πρέσβη του Μεξικού που μίλησε για μια ένα μνημειώδη εορτασμό εδώ, ε, ένας ε, υπέροχος τρόπος να συμμετέχει και το κοινό και όπως είπε και η κυρία Φιτζέραλ όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν και στο Παρίσι θα γίνει ένα φεστιβάλ πολιτισμών και αυτό που θα θέλαμε επίση και στο Μεξικό είναι απλώ να κάνουμε διαλέξει, αλλά να υπάρχει και ένα εορταστικό χαρακτήρα, ο κόσμο να, συμμετέ, να συμμετάσχει, να συγκινηθεί, να συμμετέχει και συναισθηματικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν δεν το πετύχουμε αυτό, θα έχουμε αποτύχει σε κάτι. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δώσουμε ένα διαφορετικό χαρακτήρα ε, σε όλα αυτά από ό,τι συνήθως. άλλα σχόλια. Συμφωνώ με τα σχόλια ε, που ακούσαμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη δέσμευση που δείχνετε. Και τι άλλο. Ψάχνω. Ένα θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ. Πώς μπορούμε λοιπόν να κάνουμε να συμμετάσχουν και οι μετανάστριες. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους στόχους ε, των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και της Ατζέντα 2030, κανένας να μην είναι πίσω. Εδώ είναι που συναντάνε και την Ατζέντα του Πεκίνου στην 25, ότι όλοι θα πρέπει να συμμετάσχουν και ότι θα πρέπει να ακούσουμε τις φωνές όλων. Και πάλι σας ευχαριστώ για τη σημερινή συνεδρίαση. Ε, ξεπέρασα λίγο το χρόνο μου, αλλά βλέπω ότι είστε ιδιαίτερα ενθουσιώδης για το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και πάλι. Much, uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς πρέπει να κοιτάμε το χρόνο μας. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε, γιατί αναφέρετε και νέες πτυχές. Απλά θέλω να σας ζητήσω να είστε όσο γίνεται πιο σύντομοι. Παρακαλώ, κύριε Πρέσβη. Πολύ σύντομα να σας ευχαριστήσω και πάλι για αυτήν εδώ τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας σχόλια και ιδέες. Αισθάνομαι το θέμα. Το ίδιο, ότι θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο χρόνο. Αυτό που προτείνω είναι να συνεχίσουμε τις επαφές για να δούμε κα... πώς θα προχωρήσουμε μαζί με τους ευρωβουλευτές την Επιτροπή σας και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ώστε να πραγματικά να μπορέσουμε έτσι να διαμορφώσουμε μια συμμαχία για δράση. Η ισότητα των φύλων δεν είναι ακόμα ένα θέμα. Είναι στην καρδιά της βιώσιμης ανάπτυξης και είναι στην καρδιά της Ατζέντα 2030 και πρέπει ήδη το, από το 20 να κάνουμε κάτι. Έχουμε μια ευκαιρία όχι μόνο για επαιτίους αλλά ε, για ε, δράση. Το πρώτο βήμα είναι το Μεξικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκκληση για υψηλότερη πολιτική ηγεσία. Πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Η κοινωνία των πολιτών είναι ουσιαστική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι, πρωτε, είναι πρωταγωνιστής ε, να υπάρξει λοιπόν συνεργασία με όλα τα κοινοβούλια του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλιά σας και το πώς να συνεργαστούμε με την Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας πω ότι στην περίπτωση του Μεξικού φαίνεται να ε, ε, ασκεί φεμινιστική εξωτερική πολιτική. Ευχαριστώ και το εκτιμούμε. Είναι πολύ ισχυρή συνεργασία για την χειραφέτηση των γυναικών, για δούμε ε, δηλαδή με την Κομισιόν συγκεκριμένους δρόμους συνεργασίας. Για να ενθαρρύνουμε επίσης και να στηρίξουμε τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. και να ευχαριστήσω όλους τους ε, συνεργαζόμενους. Ε, μου είπατε να είμαι σύντομος. Ακόμα μια φορά λοιπόν όμως να σας ευχαριστήσω για αυτή τη σημερινή ευκαιρία και προσβλέπω στη στενή συνεργασία μαζί σας και με τα άλλα μέλη της Επιτροπής και όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό μας το θέμα. Ναι, είναι το σημείο κίνησης μιας συνεργασίας, στενής συνεργασίας λέει η Πρόεδρος. Παρακαλώ τώρα ε, ε, πρέσβης της Γαλλίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπε με εξαιρετικό τρόπο η εκπρόσωπος της ε, ΟΗΕ ε, γυναίκες και ο πρέσβης του Μεξικό. Το μήνυμα που θα πρέπει να δώσουμε στις κυβερνήσεις μας είναι αυτό της κινητοποίησης, ώστε στις αντιπροσωπείες τους να υπάρχει η διαφοροποίηση και να εκπροσωπείται ε, ισχυρά η κοινωνία των πολιτών. Από τη δική μας πλευρά στο Παρίσι και το ίδιο συμβαίνει και στο Μεξικό θα περιμένουμε πολύ κόσμο και ελπίζουμε αυτό να επαληθευτεί. Ευχαριστώ. Thank you very much. Please. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ κυρία Μαρινάκη, σας ευχαριστώ πολύ και από τη δική μου πλευρά ένα σύντομο ευχαριστώ για όλους τους συμμετέχοντες και για την πρωτοβουλία του Ευρωκοινοβουλίου και της Επιτροπής ΦΑΜ να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος. Θα ήθελα να τονίσω τη ΣΜΚΙΟ και τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών από τη δική μας πλευρά γιατί βασικά οι δράσει μιλάνε πολύ πιο ε, ε, ηχηρά από ό,τι τα λόγια. Αποφασίσαμε λοιπόν και ο πρώτος δημόσιος λόγος της είπα, του είπα του εκπροσώπου ακριβώς πριν δύο μέρες στο φόρουμ των, των ΜΚΟ που οργανώνεται ετησίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν να υπογραμμίσει την δέσμευσή του σε προσωπικό και θεσμικό επίπεδο της Ένωσης στη στήριξη των ΜΚΟ, της κοινωνίας των πολιτών και πιο συγκεκριμένα και με μεγαλύτερη ευαισθησία υποστηρίζοντας τους, τους ακτιβιστές κάθε είδους ε, όπως ε, ε, τους ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τις γυναίκες με ύφαση στο περιβάλλον και το μέλλον του πλανήτη μας. Όλοι μας λοιπόν υποστηρίζουμε <clears throat> τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ για τα πολύ ισχυρά σας μηνύματα. Όσο μεγαλύτερη είναι η προσδρόμηση των δικαιωμάτων, τόσο πιο έντονα θα πρέπει να είναι τα μηνύματα, τα δικά μας, ε, πρακτικά μέτρα, δραστικά μέτρα υπέρ τη ισότητας. Ευχαριστώ για την προπαρασκευαστική εργασία και προσβλέπουμε σε αυτή τη συνεργασία και φαίνεται ότι το 2020 θα είναι ένα πολύ ισχυρό έτος όσον αφορά την ισότητα των φύλων σε ολόκληρη την υφήλιο. Οπότε θα προσπαθήσουμε και εμείς να συμβάλλουμε στεναρά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Επιτροπή των Γυναικών και από ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ και ε, έτσι ολοκληρώθηκε η εξέταση αυτού του σημείου της ημερησίας διάταξης. Και Τώρα θέλω να σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, γιατί εμείς θα προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Thank you.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 Ähm, Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, 10 και 11, το είχα ανακοινώσει και προηγουμένως. Θα τα δούμε από κοινού, γι' αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Francis Fitzgerald. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους για τις θετικές τους απαντήσεις ε, και τις τροπολογίες, στην επικοδομητική δουλειά. Έχουμε καλή βάση για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας. Για τις δύο απαλλαγές, ε, ευχαριστώ τον κόσμο για τη δουλειά του Για την απαλλαγή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε 26 τροπολογίες στην έκθεση και γι' αυτό έχουμε προτείνει πέντε συμβιβαστικέ. Οι συμβιβαστικέ 1, 3 και 5 θέλουν να ενισχύσουν την ευθυγράμμιση τη διασταση των φύλων και τον συνυπολογισμό στην κατάρτιση του προπολογισμού σε όλη τη διάρκεια τη δημοσιονομική διαδικασία και για το μελλοντικό ποδοπού. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό σημείο. Ε, πολλοί το τόνισαν αυτό. Επιπλέον, οι 1, 4 και 6 ε, θέλουν επιπλέον δικτέ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προπολογισμού επίση οι δύο, ε, ζητά περισσότερα για του στόχου του Ντάφνη. Άλλε τροπολογίε ζητούν ε, μια λεπτομερή εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να λάβουμε υπόψη την εξάντε αιρεσιμότητα και το κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι δείκτε ώστε να δίνεται η χρηματοδότηση. Επίση, θα πρέπει και στα εξωτερικά προγράμματα να συμπεριλαμβάνεται η διάσταση του φύλου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο των πρόσφατων συζητήσεών μα και των εργαλείων. Και θα πρέπει να υπάρξουν σχέσει συνεργασία μεταξύ των εξωτερικών και των εσωτερικών προγραμμάτων για να διευκολύνουμε τα εθνικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε του στόχου ότι των φυλών. Η ισότητα των φύλων πρέπει να ληφθεί υπόψη και στην μετανάστευση και τι πολιτικέ ασύλου. Ε, και τέλο, μια ανανεωμένη έκκληση για μια στρατηγική ισότητα των φύλων. Εδώ αναπομονώ για τα σχόλιά σα Τώρα για την απαλλαγή ε, την επόμενη έχουμε Επίση, τροπολογίε στην ευθυγράμμιση τη ισότητα σε όλε τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δύο σημειώνει τη συνεισφορά που έκανα και εγώ προηγουμένω στην Επιτροπή των Γυναικών, στηρίζει τη δουλειά μα και στην τρία. Υπάρχουν σχολεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλε τι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, όχι μόνο τη δική μα. Άλλε τροπολογίε περιλαμβάνουν εκκλήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Συνέδριο να ασχοληθούν με τη δυνάμει τη διάσταση των φύλων. Ε, πράγματα που έχουν γίνει στην όλη διαδικασία, την νομοθετική και του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ληφθούν υπόψη. Και σημειώνω τι τροπολογίε που ε, αναφέρονται στη δράση του ΙΓΚΕ ω εργοδότη. Θα πρέπει να δούμε τι απόψει των συναδέλφων και θα ρωτήσω ενδεχομένω του συναδέλφου περαιτέρω διευκρινιστικέ για να δω τι θέλουν να περιληφθεί στι τροπολογίε. Θα συνεννοηθούμε διμερώ στη συνέχεια, εφόσον χρειαστεί. Για τι δύο εκθέσει, θα ήθελα να πω πολύ σύντομα ότι για τι τροπολογίε που θέλουν να αλλάξουν τον όρο gender σε sex, φίλο σε φίλο, θα ήθελα να μην αλλάξει. Μιλάμε για ισότητα των φύλων, gender equality και θα συνεχίσω να το λέω έτσι. Θέλω να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές για την ε, ε, επικοδομητική του συνεργασία και ελπίζω να περατωθούν οι εκθέσεις για να ψηφιστούν τον Γενάρη. Ε, ακόμα είμαστε σε πορεία ε, εξέλιξη των εκθέσεων. Ευχαριστούμε και τώρα και εισηγητές, η κυρία Βίλια Μπλίνκεβιτσιούτε για του σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την κοινή μας δουλειά, για την καλή μας συνεργασία. Ως σκιώδης εισηγήτρια για τον προπολισμό του 2018 έχω υποβάλει και εγώ τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φίλων που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε όλε τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευθυγράμμιση. Διότι η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι θεμελιώδη αξία. Επίση, εξ όσων καταλαβαίνουν, η συγκέντρια συμφωνεί και θα τα συμπεριλάβει στις συμβαστικές της. Κατά τα άλλα, να πω ότι ο προπολογισμό δεν είναι εξαίρεση εδώ. Και η ευθυγράμμιση της, ισότητα, της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας είναι κάτι σημαντικό. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε ίση πρόσβαση για όλους στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τα προγράμματά της και την συμμετοχή των γυναικών στα προγράμματα αυτά. Νομίζω η ισότητα των φίλων πρέπει να αναφορθεί όλος ιδιαίτερος. Εδώ πρέπει να βρούμε μια κατάλληλη δημοσιονομική γραμμή που να στηρίζει την ισότητα των φίλων και τα γυναικεία δικαιώματα. Όσο για το πρόγραμμα Δάφνη, η μειωμένη χρηματοδότηση του προγράμματος ε, είναι επίση ένα σημαντικό σημείο. Είχαμε προβεί σε κοινή δήλωση για το θέμα αυτό και για. Εδώ λοιπόν ε, και γι' αυτό πρέπει να γίνει κάτι στα πλαίσια της ευθυγράμμισης, της διάστασης, της ισότητας των φύλων, όσο σχέση με όσα έγιναν την τελευταία αιτία. Ε, θα πρέπει να έχουμε μια σαφή θέση στην Επιτροπή μας, Εξ όσων καταλαβαίνω, η εισηγήτρια έχει ήδη υποβάλει πέντε συμβαστικέ λύσεις. Θα τις περάσουμε από την εξέτασή μας, για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε τελικώς και στην Επιτροπή μας όσο για τον προπολογισμό του Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων. Έχω επίσης υποβάλει μια σειρά από σχόλια και θέλω να τονίσω ξανά ότι ο ρόλος του Ινστιτούτου είναι πολύ σημαντικός για το πώς εξετάζονται διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας ε, κτλ. Πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες του Ινστιτούτου για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα. Πιστεύω ότι πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχει μόνο η Επιτροπή ΦΑΜ αλλά και οι υπόλοιπε κοινοβουλευτικέ βιοτροπέ του Κοινοβουλίου συμμετέχουν σε αυτέ τι δραστηριότητε. Και θα πρέπει και εμείς να υποστηρίξουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Εδώ θα πρέπει το Ινστιτούτο να παίρνει αρκετή χρηματοδότηση, ώστε να μπορεί να προσλαμβάνει ε, τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους. Αλλιώ θα υπάρξουν αρνητικέ εξελίξει. Αυτές είναι οι προτάσεις μου και η εισηγήτρια ανέφερε τρεις συμβιβαστικέ. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε πολλά σημεία σύγκληση για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Τουρέτ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Φιτζέραλτ και όλους τους κοιόδης για το ποιοτικό τους ε, έργο πάνω σε αυτές τις δύο απαλλαγές για το 2018, τι αφορά την ΑΕΓΕ είτε τον Γενικό Προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι τρεις συμβιβαστικές τροπολογίες ε, είναι απόλυτα ικανοποιητικέ, λαμβάνουν υπόψη τις τροποποιήσεις που πρότειναν οι διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Για άλλη μια φορά λοιπόν, Φράνσις, ευχαριστούμε πολύ. Όσον αφορά την ΑΕΓΕ, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, η δουλειά μας εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική, η δουλειά όλων μας σε αυτή την Επιτροπή, διότι πρέπει να προωθήσουμε τις εργασίες ε, και της Κομισιόν, ούτω ώστε με οριζόντιο τρόπο να προωθήσουμε την ατζέντα, να ξέρουμε ποια είναι τα νούμερα, να ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Οι στατιστικές της ΆΕΚΕ είναι για μας πάρα πολύ σημαντικές, για όλους εμάς που λαμβάνουμε αποφάσεις, αλλά και για όλους τους πολίτες, των οποίων η ενημέρωση είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας. Είναι λοιπόν ε, πρωταρχική σημασία να έχει το ΆΕΓΕ ε, και ε, στελέχη και ανθρώπινο δυναμικό αλλά και οικονομικούς πόρους για να μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους μας. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να συμπεριλάβει λοιπόν όλα αυτά στον στην κατάρτιση του προϋπολογισμού όσον αφορά τώρα το γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό και πάλι να εντάξουμε τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης, αλλά και στην ε, εφαρμογή και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Δηλαδή, και κατά την κατάρτιση του προπολογισμού και κατά την εκτελέσή του και κατά την αξιολογησή του θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τη διάσταση του φύλου. Θα πρέπει να είναι μια προτεραιότητα την οποία να παρακολουθούμε συνεχώ στο πλαίσιο του ενωσιακού προπολογισμού. Να προωθούμε δηλαδή την ισότητα των φύλων. Και γι' αυτό έχουμε ανάγκη στοχευμένες δράσεις για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους σχετικά με την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Θα πρέπει επίσης να δίνουμε ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί θεωρώ απαράδεκτο τη σήμερον ημέρα 2019 προγράμματα όπως το Erasmus Sin ή η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων να έχουν τόσο χαμηλή γυναικεία συμμετοχή. Θα πρέπει επίσης το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων να συμπεριλάβει τη διάσταση του φύλου. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να προσμετρώνται στους δείκτες απόδοσης του προϋπολογισμού, να έχουμε στόχους ε, οι οποίοι να είναι αριθμητικοί, ε, γιατί με αυτόν τον τρόπο μόνο τότε θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τους στόχους μας και να τους επιτύχουμε. Ευχαριστούμε εκ μέρους των Πρασίνων η Μόνικα Βάν, αλλά νομίζω δεν είναι εδώ. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν ε, άλλες πολιτικές ομάδες που θέλουν να πάρουν το λόγο. ID, ECR, κανείς που θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Ολοκληρώνουμε λοιπόν ε, με τις ε, τροπολογίες. Θέλετε να ξαναπάρετε το λόγο. Όχι, εντάξει. Ευχαριστώ λοιπόν όλους για τη συμβολή σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό το σημείο ε, της ημερήσιας και πηγαίνουμε στο σημείο 9, ιδιαίτερα ενδιαφέρον, η παρουσίαση εκ μέρους της ΆΕΓΕ, του Ευρωπαϊκού Ιστιντούτου για την Ισότητα των Φύλων. Και τώρα η κυρία Λάγκμπακ έχει τον λόγο. Έρχεται, την καλωσορίζουμε είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την παρουσίαση στην ε, διάσκεψη που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Και θέλουμε λοιπόν να μάθουμε τα αποτελέσματα των εργασιών σας, ε, κάποια καλύτερα, κάποια ίσως λιγότερα. Έχετε το λόγο λοιπόν για να κάνετε την παρουσίαση και στη συνέχεια θα διεξάγουμε μια συζήτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα-πρώτα, χαίρομαι ιδιαίτερα. Είναι η πρώτη φορά και ίσως η τελευταία που βρίσκομαι εδώ στην ε, Επιτροπή ΦΑΜ. Είναι λοιπόν η ΆΙΓΕ ένα πολύ σημαντικό, παρέχει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη της, του θεματολογίου. Ε, αυτά όμως θα σας τα πω και στη συνέχεια. Άκουσα ένα μέρος ε, της συζήτησης για την απαλλαγή. Ε, θίξατε και το θέμα των εργαζομένων στην ΑΕΓΕ. Ευχαρίστω να σας πληροφορήσω, διότι όχι μόνο σχετίστε με τις ιδιαιτερότητες ε, του Ιστιντούτο μας, αλλά και με τους γενικότερους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα θέμα που δεν αφορά λοιπόν μόνο την ΑΕΓΕ. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν, ε, τι κάνουμε, νομίζω ότι κάποιοι ήδη ξέρετε εδώ στην Επιτροπή και γενικότερα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, θα σας κάνω μια πολύ σύντομη ενημέρωση όμως παρόλα αυτά ε, στο πώς, συνεργαζόμαστε, πώς εργαζόμαστε για να στηρίζουμε εσάς, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο και όλη την κοινωνία των πολιτών βεβαίως. Έχουμε λοιπόν ένα πεδίο έρευνας και έχουμε τον δίκτυ ισότητας. Να σας το δείχνω, αλλά βλέπω ότι έχετε κι εσείς ε, ένα αντίτυπο. Ε, είχε προταθεί από την προηγούμενη νομοθετική περίοδο να υπάρξει ένα τέτοιο εργαλείο ε, παρακολούθησης και θα σας πω με λεπτομέρειες στη συνέχεια περί τίνος πρόκειται. Όμως η διοίκηση του Ινστιτούτου ενέκρινε αυτός ο δείκτης να υπάρχει και να γίνεται κάθε χρόνο. Δεν έχουμε πολλούς πόρους, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να διαπιστώνουμε ότι κάποιος χάρος πάνε προς τα πάνω, κάποιος άλλος προς τα κάτω και είναι πολύ σημαντικά, ε, σημαντικοί οι δείκτες αυτοί για να δίνουν το ε, μήνυμα στις κυβερνήσεις του τι να κάνουν. Ε, επίσης μπορούμε να επικεντρωθούμε σε κάποια συγκεκριμένα θέματα με αυτόν τον τρόπο. Ε, του χρόνου λοιπόν θα επικεντρωθούμε περισσότερο στην υγεία. Μέχρι τώρα ε, είχαμε επικεντρωθεί στην ισότητα των φύλων. Και εσείς το αναφέρετε και στην απαλλαγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή ΦΑΜ επί τη βάση των ευρημάτων μας να συμπεριλαμβάνει σε όλους τους τομείς πολιτικής τη διάσταση του φύλου. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι η έκθεση του Πεκίνου Ξέρετε ότι ε, ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια, γίνεται μια αξιολόγηση της διεθνούς δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το πώς συμμετέχει, για παράδειγμα, στις διεθνείς συμβάσεις με τον τα κτλ. Γι' αυτό είχε γίνει και η πλατφόρμα του Πεκίνου. Για να δούμε λοιπόν πώς συμβάλλει κάθε χώρα. Σε 10 ε, χρόνια όμως όπως σήμερα θα έχουμε, το κάνουμε ήδη και θα ενοποιούμε περισσότερο τις, ε, τα συμπεράσματα ανά χώρα. Επίσης, ε, αυτό που τονίστηκε στην διάλεξη για τον δίκτυ ήταν ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε μια ενιαία παρακολούθηση. ξέρουμε τι γίνεται, αλλά πώς το κάθε κράτος εφαρμόζει αυτά τα στοιχεία. Δεν υπήρχε παρακολούθηση, δεν ξέραμε. Νομίζουμε λοιπόν ότι και αυτό θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στη νέα στρατηγική της ε, ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι άλλο επίσης. Έχουμε μια βάση δεδομένων με στατιστικές για την ισότητα των φύλων και θα πρέπει, θα είναι, είναι ήδη μάλλον αυτή προσβάσιμη από κάθε ευρωβουλευτή και σας καλώ να κάνετε πραγματικά χρήση της βάσης δεδομένων μας, την οποία επικαιροποιούμε τακτικά. Επίσης, έχουμε ε, την συμπερίληψη της διάστασης του φύλου. Όχι μόνο γενικά, ε, στους διάφορους τομείς πολιτικής, αλλά έχουμε και την συμπερίληψη της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού. Όλα αυτά τα έχουμε στην πλατφόρμα μας ε, στο διαδίκτυο. Ε, πριν από κάποια χρόνια ξεκινήσαμε μια τομεακή προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ε, για παράδειγμα, αν θέλετε να μάθετε πώς η αλλήλεια συνδέεται με την ισότητα των φίλων, μπορείτε να πάτε στο site και να δείτε, γιατί παρουσιάζουμε τα επιχειρήματα και λέμε να, τι πρέπει να γίνει για να πάμε πιο πέρα. Και αυτό είναι σημαντικό για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Συμμετέχουμε ε, λοιπόν στην ε, συμπερίληψη της διάστασης του φίλου, στην ε, κατάρτιση του πολυπολογισμού. Το κάναμε και την Ρουμερική Προεδρία, ε, συζητήθηκε το θέμα και οι Υπουργοί Απασχόλησης τώρα προωθούν το θέμα. Έχουμε επίσης αναλύσει ε, τους πόρους που δεχόμαστε. 1% για την ισότητα των φύλων δεν είναι αρκετό, αυτό είναι σίγουρο. Θα πρέπει λοιπόν ε, οι κύριες δράσεις μας ε, για την ισότητα των φύλων ε, να μεταφραστούν επίσης και σε κατάλληλη χρηματοδότηση. Του χρόνου λοιπόν θα δούμε τις δημόσιες συμβάσεις περισσότερο όσον αφορά τη διάσταση του φύλου και πάλι. Η βία τώρα κατά των γυναικών στον δίκτυ δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μία ανάλυση όσον αφορά την ε, ε, εμπορία ανθρώπων, γυναικών. Ξέρετε ότι είναι οι γυναίκες που πλήττονται κυρίως από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά δεν έχουμε αρκετά δεδομένα. Έχουμε όμως συνεργαστεί με τις δικαστικές αρχές, την αστυνομία, ψάξαμε μάρτυρες, αναζητούμε μάρτυρες, ήδη, δηλαδή ο ίδιος ο κόσμος να ε, συμμετέχει προσφέροντας στοιχεία, να υπάρξει ε, τα θύματα τα ίδια, να κάνουν ε, καταγγελία και να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση του θέματος. Θα ήθελα λοιπόν τώρα σήμερα να σας ε, δείξω κάτι που υπάρχουμε ήδη ξεκινήσει στο διαδίκτυο. Έχουμε αναπτύξει και έχουμε ολοκληρώσει ε, στο πλαίσιο της διεθνούς ε, διακοινοβουλευτικής συνεργασίας ένα ερωτηματολόγιο για να κάνουμε μια αυτοαξιολόγηση. Είναι ένα εργαλείο για οποιοδήποτε κοινοβούλιο για να μπορέσει να αξιολογήσει πώς ε, οι ευκαιρίες αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με τις εθνικές, τις περιφερειακές αρχές, τα τοπικά κοινοβούλια, πώς μπορούν όλα αυτά να αξιολογηθούν. Υπάρχουν δύο υπηρεσίες. Η μία πηγαίνει σε βάθος, και μας δίνει πολύ καλές πληροφορίες για το πού υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και η άλλη είναι μια πιο γενική προσέγγιση που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες. Και εδώ σας παρουσιάζουμε κάποια στοιχεία. Βλέπετε πώς λοιπόν διαφέρουν τα πράγματα ανατομέα, πώς αλλάζουν. Αλλά για παράδειγμα, όταν θέλουμε να δούμε πόσες γυναίκες μπαίνουν ε, στα κοινοβούλια όχι μόνο βουλευτές, αλλά και διοικητικό προσωπικό τότε διαπιστώνουμε πόσο έχουμε προχωρήσει εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και πώς τα πράγματα εδώ είναι καλύτερα από ότι ο διεθνής μέσος όρος. Μετά αν κοιτάξουμε το νομοθετικό μέρος, ε, τις φυλαξη φύλαξης παιδιών, του παιδικού σταθμού, πώς όλα αυτά συμβάλλουν ε, στην ισότητα των φύλων, πώς σχετίζονται όλα αυτά. Ε, θα σας δείξω εδώ κάποια στοιχεία αυτού του δίκτυ. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω πώς ακριβώς ε, δουλεύει, αλλά αν ανοίξετε την ιστοσελίδα μας, θα διαπιστώσετε ότι έχουμε έχουμε πέντε mm-hmm. δείκτες για πέντε διαφορετικούς τομείς mm-hmm. που δείχνουν ε, σε ποιο βαθμό βρισκόμαστε πάνω από το κατώτατο όριο. Αυτό είναι το πράσινο. Το κίτρινο είναι που υπάρχουν ακόμα κίνδυνοι και μετά υπάρχει το κόκκινο που είναι ε, οι πιο ευαίσθητες περιοχές. Έχουμε λοιπόν ε, αξιολογήσει όλες τις εθνικές, τα εθνικά κοινοβούλια. Έχουμε ρωτήσει, για παράδειγμα, τις γυναίκες κατά πόσο αισθάνονται ασφαλείς ε, όσον αφορά τον ε, εκφοβισμό κτλ. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορείτε να το βρείτε στο, ε, στην ιστοσελίδα μας. Επίσης, ε, συνεργαζόμαστε και με την ΚΟΖΑΚ όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια και έχουμε επισημάνει ότι όλα τα κοινοβούλια με κόκκινο θα πρέπει να γίνουν πράσινο. Εδώ ε, είχαμε πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις και φέτος ο δείκτης έχει επικεντρωθεί στην εξισορρόπηση επαγγελματικού οικογενειακού βίου. Ξέρετε ότι είναι ένα θέμα που είναι πολύ έμφυλο, αφορά ιδιαίτερα τα φύλλα για τη ζωή μας, γυναίκες που δουλεύουν. Ε, αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπήρξε συγκεκριμένο αίτημα της ε, πρώην Επιτρόπου για την Ισότητα των Φίλων, τη κυρία Γιούροβα, για να δημιουργήσουμε ένα βαθμολόγιο για την εξισορρόπηση οικογενειακού επαγγελματικού βίου. Ψάξαμε νέε εναλλακτικέ προσεγγίσει για το βαθμολόγιο αυτό, ώστε να υπάρξει μια σωστή εξισορρόπηση για πολλέ διαστάσει που δεν έχουν ληφθεί ω τώρα παρκώ υπόψη και πρέπει να τονιστούν. Τι κάνουμε λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τα βλέπετε ανάλογα με το κάθε ποσοστό πώς έχουν εξελιχθεί από το 2005 και βλέπουμε ότι το 2005 υπάρχουν πολύ ε, μικρή αύξηση, τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε πέντε χρόνια. Ε, και και να ξέρουμε σε ποιους τομείς έχουμε πάει πολύ γρήγορα και ποιους όχι. Ε, όπως κάποιος είπε σήμερα, το 2019 είναι απαράδεκτο να είναι ακόμα εκεί τα δεδομένα. Και εμεί έτσι λέμε, είναι απαράδεκτο να έχουμε τόσο αργή πρόοδο. Μετά, αν δούμε τι ε, μεμονωμένε ε, επιδόσει των κρατομελών, βλέπετε η Σουηδία από την αρχή ήταν ε, πρώτη των πρώτων, μετά η Δανία και η Γαλλία. Σε άλλα κράτη-μέλη λοιπόν είχαμε επιδόσει καλύτερε από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι πολλοί αυτοί που είναι κάτω, στην Πορτογαλία α πούμε. Πολύ καλή εξέλιξη. 3,9 για την Πορτογαλία. Και κυρίω ε, πολιτική, στη δικασία πολιτικών αποφάσεων. Στην Εσθονία. Στον τομέα ε, γνώση, χρήμα και εξουσία. Εδώ λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε να δώσουμε περισσότερη δυνατότητα στις βουλές, γιατί υπάρχει περιθώριο ε, για βελτίωση. Βλέπουμε, ας πούμε, να είναι έκτη Λιθουανία, ενώ που ήταν... Ε, αλλού τα, ε, τα πράγματα Και κυρίω όλα έχουν ε, παρουσιάσει βελτίωση γιατί οι γυναίκε συμπληρωμάτων στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Δείτε λοιπόν συγκεκριμένου τομεί. Βλέπουμε ότι το θέμα είναι η εξουσία. Εκεί έχουμε ε, την πιο γοργή ανάπτυξη, αλλά με χαμηλό ποσοστό. Και μετά ο χρόνο. Ο χρόνο που έχει σχέση με την εξισορρόπηση. Θα σα δείξω μετά πώ αναλύσαμε τα στοιχεία. Υγεία και χρήμα Εκεί βλέπετε να υπάρχουν οι περισσότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ξέρετε πώς είναι το πλαίσιο και οι ποσοστώσεις. Τα έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Τι έγινε ε, με, το άλμα στις ποσοστώσεις, εκεί όπου προβλέφθηκε πολιτικός και νομικός ε, η ποσόστοση άνδρες και γυναίκες αναγκαστικά στην ίδια ποσόστοση. Εκεί τα πράγματα γνώρισαν εκρηκτική πρόοδο. Ε, τώρα το βαθμολόγιο έχουμε μονομένους δείκτες, έχουμε την ε, μακροπρόθεσμη φροντίδα, την ε, φροντίδα των παιδιών, την επαγγελματική κατάρτιση. Κοιτάμε λοιπόν με διάφορους δείκτες και μετά ε, έχουμε αναλύσει τις δύο διαστάσεις της φροντίδας και μετά την επαγγελματική κατάρτιση μαζί με την ε, εκπαίδευση. Πρέπει να κοιτάξουμε ποια επαγγελματικά Ινστιτούτα παρέχουν τις γονικές άδειες και τι υποδομές διαθέτουν. Είναι κάτι καινούριο υποδομές, αλλά πρέπει να ε, το δούμε προσεκτικότερα. Βρήκαμε κάποια μοτίβα που λειτουργούν με βάση τη διάσταση του φύλλου και πρέπει να το μελετήσουμε καλύτερα. Για τις γονικές άδειες τώρα, τι βλέπουμε. Βλέπουμε τρία μόνο από τα νέα κράτη-μέλη. Οι γυναίκες και οι άνδρες με παιδιά να έχουν τη δυνατότητα, όλοι οι γυναίκες και οι άνδρες, να πάρουν γονική άδεια. Τα τρία αυτά κράτη-μέλη είναι η Εσθονία, η Φινλανδία και η Σουηδία. Οι υπόλοιποι σε ένα βαθμό έχουν τις δυνατότητες, αλλά υπάρχουν και περιορισμοί. Βλέπετε τις 18. Αυτά έχουν να κάνουν και με τις συνθήκες απασχόλησης. Μιλάμε για αυτοαπασχολουμένους. Εκεί δεν μπορούν να πάρουν γονική άδεια. Βλέπετε σε ποια χώρα και τα ζεύγη σύντροφοι φίλου. Εκεί δεν παίρνουν γονική άδεια. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τα αίτια. Βλέπουμε το σημαντικότερο αίτιο για να μην μπορεί κάποιο να πάρει γονική άδεια. Η ανεργία και η έλλειψη επαγγελματική δραστηριότητας. Βλέπουμε ότι περισσότερο εδώ στην ανεργία έχουμε γυναίκες Και μετά οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άντρες. Οι γυναίκες είναι περισσότερο ανεργές και είναι και μεγαλύτερα θύματα εφόσον είναι αυτοαπασχολούμενες. Εδώ μιλάμε για τι υπηρεσίε φροντίδα, αυτοαπασχολουμένου. Ε, άρα ο κίνδυνο είναι μεγαλύτερο για του άντρε. Εκεί και μετά έχουμε και τα χαρακτηριστικά ένα νοικοκυριό. Έχουμε 10 ε, κράτη-μέλη, όπου για τα ζεύγη δύο φύλου δεν είναι επιλέξιμη. Με τι νέε συμβάσει, με όλη τη συζήτηση για την ψηφιοποίηση, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία μπορούν να εξεταστούν στα πλαίσια τη νέα στρατηγική, αλλά και στι διάφορε οδηγίε που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό εξέταση από τη Νέα Επιτροπή. Επίσης, για τη συγκεκριμένα στοιχεία των ε, ε, υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών. Βλέπουμε ότι η διάσταση αυτή είναι ένα πολύ σημαντικό κριτήριο για να αλλάξει κάτι στη ζωή των γυναικών. Όταν είναι επιδοτούμενη η φροντίδα αυτή, αυτό είναι τεράστιο τεράστιο στοιχείο που συμβάλλει στη μείωση της ανισότητας. Βλέπουμε οι στόχοι της Βαρκελόνης να είναι αυτοί που επιδιώκουμε από 9 χρόνια. 9 χρόνια αργότερα βλέπετε το πράσινο κύκλο. Δεξιά 11 κρατημέλη όπου έχουν επιτευχθεί και δύο στόχοι. Στον κίτρινο έχουμε 10 κρατημέλη που κάποιοι στόχοι επιτεύχθηκαν και κάποιοι έτσι και έτσι. Και μετά έχουμε τον κόκκινο κύκλο, αυτοί που δεν έκαναν τίποτα. Και να σας δείξω και το τελευταίο. Πώς αναλύουμε την ισότητα των φύλων, τον μέσο όρο ισότητας των φύλων και πώς αυτό συνδέεται με την φροντίδα των παιδιών την διάθεση φροντίδας. Δεν θα εκπλαγείτε οι χώρες που είναι στη γωνία, στα δεξιά, Σουηδία είναι η πρώτη των πρώτων. Μετά είναι η Δανία, κάτω χώρες, Λουξεμβούργο, Βέλγιο και Γαλλία. Με κάποιες διαφορετικές επιδόσεις στην κλίμακα της ισότητας των φύλων, βλέπουμε ότι η ισότητα των φύλων πραγματικά πάει χέρι-χέρι με τις εξελίξεις στην φροντίδα των παιδιών. Αυτά είναι λίγο πολύ τα στοιχεία. Ξέρω δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, οπότε καλύτερα να κρατήσουμε και λίγο χρόνο για ερωταπαντήσεις. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά που μας είπατε πραγματικά προκαλούν εκατοντάδες ερωτήσεις στο μυαλό του καθενός. Ευχαριστούμε για τη δουλειά σας και για τη δουλειά που κάνει το ΕΓΚΕ για ε, όλους τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες. Η Μαρία Μανουέλ είναι η πρώτη που ζήτησε το λόγο. Και εγώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλο αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει, γιατί χωρίς ε, στοιχεία δεν μπορούμε να διατυπώσουμε πολιτικές που να έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την αναφορά που κάνατε στη χώρα μου στην πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μου. Εγώ ήμουν υπουργό αρμόδια και πραγματικά με συγκινήσατε με τα καλά σας λόγια. Κάναμε πολλά και γι' αυτό στην Πορτογαλία τώρα είμαστε σε μια σχετικά, σχετικά καλή κατάσταση. Έχουμε λοιπόν τώρα τέσσερι επιλογέ. Πρέπει να προσέξουμε τα στοιχεία για την οικιακή βία, τα οποία είναι λυπή και συλλέγονται με διαφορετικά κριτήρια στι διάφορες χώρε τη Ένωση και εν γέννη πρόκειται για στοιχεία τα οποία δεν είναι πολύ αξιόπιστα. Δεύτερον, έχουμε στοιχεία για τι ε, μισολογικέ διακρίσει θα χρειαζόμαστε καλύτερα αποτελέσματα γιατί δεν ξέρουμε πού να κατευθύνουμε τις κυρίες μας προσπάθειες. Χρειαζόμαστε δηλαδή καλύτερα στοιχεία για την ε, ε, μισθολογικέ διακρίσει διακρίσεις. Το τρίτο αφορά το σημερινή υπόθεση, τη συνδυασμό μεταξύ της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά συχνά το ξεχνάμε. Και κυρίως δηλαδή πρέπει να έχουμε πιο ειδικευμένα στοιχεία. Στην Πορτογαλία το πρόγραμμα που έχουμε κάνει, τι κάνει, πιστοποιεί εταιρείε και μικρομεσαίες και τη στηρίζει με κοινοτικά χρήματα ώστε να αναπτύξουν εσωτερικά καλές πρακτικές και να έχουν μια πιστοποίηση όπως αυτή που εσείς είπατε με την ΕΖΑ 9000 και άλλες προδιαγραφές. Ήταν πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί αυτό το σύστημα πιστοποίησης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, όσον αφορά δηλαδή τις καλές πρακτικές τόσο για τους ιδιώτες, για τον ιδιωτικό τομέα όσο και για το δημόσιο τομέα που πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα και μια καλή πρωτοβουλία προέκυψε είναι μια καλή πρωτοβουλία λοιπόν, το προτείνω στην Πρόεδρο ε, για να αναλάβουμε πρωτοβουλία ώστε να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό στάνταρ για την πιστοποίηση για την ισορροπία μεταξύ προσωπική και επαγγελματική ζωή. Γιατί δεν υπάρχει ισορροπία, δεν μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε. Μπορεί να φτιάχνουμε εμεί οδηγίε για τι women on board, για τι γυναίκε στα δικτικά συμβούλια, αλλά πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα επιλογή οι γυναίκε, που δεν είναι η ίδια για άνδρε και γυναίκε. Και τέλο. Ε, προσοχή στα δεδομένα τα οποία δεν είναι ε, σωστά γιατί οι αλγόριθμοι, εάν βασιστούν σε λάθος στοιχεία, οι αλγόριθμοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα σε πολλούς πολλούς κλάδους. Και πάλι σας ευχαριστώ που είστε εδώ και που συνεργάζεστε μαζί μας για να μας δώσετε τις προποθέσεις για να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε στους αγώνες μας. Ευχαριστώ πολύ. Η ευχαριστώ πολύ για την ε, πολύ ε, καλή σας δουλειά και ευχαριστώ και την συνάδελφο ε, Μάρκες για την εξαιρετική δουλειά που έκανε στην Πορτογαλία όσο ήταν εκείνη αρμόδια υπουργό. Τη συγχαίρω θερμά. Πρέπει να πω ότι χαίρομαι πολύ που βλέπω σε αυτά τα στοιχεία κάποια στοιχεία που είναι τόσο πολύ σημαντικά, ποσοστώσεις ένα, ποσοστώσεις δουλεύουν. Αυτό δείχνουν αυτά τα στοιχεία. Έπειτα, επιδοτούμενες ε, ε, δομές φροντίδας παιδιών πέρα, ε, αντί για άλλες λύσεις. Αυτή είναι πολύ σημαντικά αποτελέσματα αυτά για, σε σχέση με τις πολιτικές που έχουν ασκηθεί. Ε, ε, ε, δεν θέλω να σχολιάσω τα δεδομένα γιατί συμφωνώ απόλυτα με το γεγονός ότι χρειαζόμαστε πολύ πιο καλά στοιχεία, ιδιαίτερα για την έμφυλη βία. Επίσης χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα για το πώς η έμφυλη βία συνδέεται με κοινωνικο-οικονομική κατάσταση γιατί εκεί υπάρχει ένα, ε, <clears throat> μια προκατάληψη που χρησιμοποιείται και από πολιτικές άποψεις, από πολιτικά κινήματα που αρνούνται την βία, αρνούνται τις ανισότητες των φύλων, αρνούνται τα θέματα του φύλου. στην Ισπανία υπήρξαν κάποια πολιτικά κόμματα πρόσφατα που είπαν ότι ναι, η ισορροπία των φύλων είναι πρόβλημα των μεταναστών μόνο, των φτωχών κτλ. Και, εν πάση περιπτώσει πρέπει να έχουμε καλύτερα στοιχεία ε, για αυτό Τέσσερι τις στοιχείες, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι... Αν δεν έχουμε σωστά στοιχεία, <clears throat> έχουμε να κάνουμε μετά με επικίνδυνες ρητορικές και επικίνδυνο λόγο. Θα πρέπει ε, να πιώσουμε επίσης τα κράτη-μέλη Πρέπει να πιέσουμε για έγκαιρες έρευνες όμως κάθε φορά. Κάποιες φορές κάποιες χώρες καθυστερούν, ε, δεν κάνουν απογραφές ας πούμε, κάθε 6 χρόνια. Δεν το κάνουν, δεν λαμβάνουν υπόψη σοβαρά αυτή την έρευνα που για τους δικούς μας σκοπούς είναι πολύ ουσιαστική. Όταν λοιπόν μικραίνει και μικραίνει το δείγμα, δεν στέκουν πια ε, οι στατιστικές. Θα αναφέρω μόνο ένα στοιχείο για να μην ακρηγορήσω πολύ, κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζουμε σωστά. Είναι κάποιες ομάδες ηλικιακέ, κυρίως οι ηλικιωμένοι, για μας όμως είναι πολύ σημαντικοί οι νέοι. Το δείγμα των νέων είναι πολύ μικρό και εκεί πραγματικά χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία, γιατί εκεί ξεκινάνε όλα. Και δεν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα αυτό που έχουμε και άρα τα στοιχεία μας. Επίσης, κοινωνικονομικά στοιχεία δεν έχουμε αρκετά. Δεν μπορούμε να κάνουμε συνδυασμούς, λοιπόν, αλλά ειδικά για τους νέους. Εξαρτάται κάποιες φορές έχουμε ε, κάθε 6 χρόνια υπογραφές ή κάθε 10 χρόνια, εξαρτάται τη χώρα. Πάντως το δείγμα είναι μικρό για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Πριν μπουν στην αγορά εργασίας, πριν από την ε, μητρότητα ή ε, την πατρότητα. Πολύ δουλειά πρέπει να γίνει, το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά <clears throat> για τα δεδομένα. Και κάτι τελευταίο, εδώ σε αυτή την έκθεση έχετε εστιάσει στην ισορροπία μεταξύ προσωπικής και ε, επαγγελματικής ζωής και κοίταζε τα στοιχεία 37, σελίδες 37-38 ότι οι γυναίκες πληρώνουν το τίμημα της μητρότητας. Ίσως θα πρέπει να περιληφθεί στην ισορροπία μεταξύ προσωπικής και ε, επαγγελματικής ζωής να συμπεριληφθεί η ε, τιμωρία της μητρότητας αλλά και το πριμ της πατρότητας γιατί λειτουργούν και τα δύο αυτά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριο Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ε, το Ιστιντούτο για την εξαίρετη δουλειά του που γνωρίζουμε εδώ και χρόνια. Οπωσδήποτε τα δεδομένα που μας παρουσιάζεται τακτικά είναι ένα εξαίρετο εργαλείο πολιτικής που μας βοηθά στην λήψη αποφάσεων. Αυτό που προκύπτει από αυτά που μας είπατε σήμερα, αυτά που είπε και η Λίνα, είναι ότι οι κυριότερες ιδέες ε, που προκύπτουν από αυτά είναι ότι οι ποσοστώσεις βοηθούν την πρόοδο. Βεβαίως τα έχουμε συζητήσει αυτό, ότι μπορούμε να κάνουμε για τη συμμετοχή, μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών. Και ε, όλα αυτά μας βοηθούν βεβαίως να λάβουμε σωστές αποφάσεις. Και πάλι Νομίζω ότι έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου πρέπει να γίνει μεγαλύτερη πρόοδος και δυστυχώς προχωρούμε αργά όσον αφορά τον δίκτυ ε, τον οποίο αναφέρατε, το δίκτυ Βεβαίω, υπάρχουν ακόμα μεγάλες διαφορές μισθολογικέ, εξισορρόπηση προσωπικής επαγγελματική ζωής, συμμετοχή των γυναικών στον χώρο εργασία κτλ. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά λοιπόν όσον αφορά την πραγματικότητα και το πώς μπορούμε να την επηρεάσουμε με λήψη αποφάσεων. Ε, πρέπει να συμπεριλάβουμε όλα αυτά και στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, κάτι που δεν γίνεται μέχρι τώρα και ακόμα και σε πολλές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να πω το εξής και να κάνω και μια ερώτηση. Θα ήθελα να πω ότι ήμουν πρώην εισηγητής ε, στην ε, έκθεση για την πρόοδο της ισότητας των φύλων και για μένα τα στοιχεία ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι φέτος έχει αναλάβει η Γκουε να συντάξει την έκθεση. Αλλά ελπίζω λοιπόν ότι θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία σας. Και μια ερώτηση. Πώς νομίζετε ότι τα δεδομένα και οι δείκτες αυτοί θα χρησιμοποιηθούν ε, στην ε, χάραξη της νέας στρατηγικής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεργάζονται μαζί σας, χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας. Διαφορετικά νομίζω ότι θα μπορούσαμε εκ μέρους αυτής της Επιτροπής να προτείνουμε στην Επιτροπή να τα χρησιμοποιήσει. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ. Βλέπω, διαβάζετε αυτά που σας δίνουμε και αυτό μας δίνει μια ηθική ικανοποίηση, διότι εμείς είμαστε πραγματικά αφοσιωμένοι στο έργο μας. Και τώρα όσον αφορά τις στατιστικές για τη βία, υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια, διαφορετικά δεδομένα σε σχέση και με την κοινωνική κατάσταση. Ναι, το ξέρουμε, το έχουμε διαπιστώσει και η δουλειά μας λοιπόν ε, προσπαθεί να ενοποιήσει κάπως τους διαφορετικούς ορισμούς. Δηλαδή σήμερα δουλεύουμε, ε, εργαζόμαστε πάνω στις γυναικοκτονίες και τον βιασμό και διαπιστώνουμε ότι οι δικαστικές αρχές και η αστυνομία σε πολλά διαφορετικά κράτη έχουν διαφορετικές μεθόδους, διαφορετικούς ορισμούς. Αυτό που θέλουμε λοιπόν να κάνουμε είναι να ε, ενοποιήσουμε, να δώσουμε μια ομοιομορφία σε αυτούς τους ορισμούς και ε, να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο μας. Δεν το έχουμε επιτύχει ακόμα, αλλά θα ε, σχεδιάζουμε να είναι μέρος του δίκτυ μας, γιατί μέσα στο δίκτυ υπάρχει αυτό το κομμάτι για τη βία. Και θέλουμε λοιπόν να έχουμε και άλλους δείκτες γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν επίγνωση του προβλήματος. Χρειαζόμαστε ακόμα κάποια χρόνια, ούτως ώστε όλα τα κράτη-μέλη να έχουν τους ίδιους ορισμούς για να μπορούμε να κάνουμε σύγκριση. Όπως ε, γνωρίζετε, εδώ και πολλοί ερευνητές έχουν, ε, χρόνια, εδώ και χρόνια πολλοί ερευνητές έχουν αναγνωρίσει ότι η βία υπάρχει σε όλα τα κράτη, σε όλα τα επίπεδα. Βεβαίως γνωρίζουμε τις αδυναμίες που επισημάνατε ότι έχουμε επιλέξει, ε, να επιλέξουμε μάλλον κάποιες ομάδες σε κάποια κράτη για να δούμε και ποιες είναι οι αδυναμίες. Ελπίζουμε ότι με τη γερμανική προεδρία λοιπόν του χρόνου θα επανέλθει το θέμα και ότι θα έχουμε νέες ιδέες επ' αυτού. Όσον αφορά την εξισορρόπηση προσωπικής επαγγελματικής ζωής και τις διακρίσεις, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η έκθεση για το Πεκίνο είναι 25 έδινε κάποιες ιδέες, παρουσίαζε κάποιες χρηστές πρακτικές. Νομίζω ότι υπάρχει ήδη στο διαδίκτυο, αν δεν έχει γίνει θα γίνει σε κάποιες εβδομάδες. Παρουσιάζει λοιπόν πολλά λεπτομερή στοιχεία που χρησιμοποιούμε για την ανάλυση των 28 κρατών μελών. Μιλήσατε για αλγόριθμους. Ομολογώ ότι είμαι λίγο μπερδεμένη γιατί του χρόνου ο δείκτης, με συγχωρείτε σας είπα κάτι που ήταν λάθος πριν, δεν θα επικεντρωθεί στην υγεία, αλλά θα επικεντρωθεί περισσότερο στην ψηφιοποίηση στο χώρο εργασίας. Και θα είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση να δούμε ποια δεδομένα έχουμε, πώς μπορούμε να τα αναλύσουμε και θα δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα που αναφέρατε. Η τεχνητή νοημοσύνη βεβαίως είναι κάτι ευρύτερο και θα πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα όσον αφορά την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, αυτό που διαπιστώσαμε στο πλαίσιο του δίκτυ αλλά και στην έκθεση του Πεκίνου είναι ότι η βία δεν είναι μόνο ενδοοικογενειακή, αλλά αφορά και κάποιες ομάδες όπως γυναίκες με αναπηρίες που πλήττονται περισσότερο και επίσης γυναίκες μετανάστριες. Είναι στην ζώνη κινδύνου. Όσον αφορά την έρευνα που προτείνατε, συμφωνώ απόλυτα. Κάτι που κάναμε και που αναφέρεται και στην ε, έκθεση του Πεκίνου ήταν η μισθολογική διαφορά. Όταν αναφέρουμε την ε, μισθολογική διαφορά και όταν λέμε ότι τώρα έχει κάπως ε, περιοριστεί, είναι γιατί ε, υπολογίζουμε μόνο την οριαία διαφορά. Όμως όταν υπολογίζουμε το σύνολο των απολαβών, τότε φαίνεται πραγματικά η μισθολογική διαφορά και τότε μπορούμε να μιλήσουμε για τα πριν που αναφέρατε ε, μητρότητας ή πατρότητας. Το 47% λοιπόν του χάσματος μισθολογικού παραδίδεται σε γυναίκες που έχουν παιδιά κάτω των 7 ετών ένα πολύ σημαντικό ποσοστό επί του οικογενειακού εισοδήματος. Πολύ σημαντικό, αξιοσημείωτο αυτό. Ε, το τίμημα που πληρώνουν οι γυναίκες για τη μητρότητα δηλαδή. Τώρα όσον αφορά την στρατηγική για τα φύλλα, βεβαίως αυτή την χαράσει η Κομισιόν και η Επίτροπος Ντάλι. Προς το παρόν δεν ε, ζήτησαν τα δεδομένα μας, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα τα χρησιμοποιήσουν. Υπάρχει και η Γενική Διεύθυνση ε, που παρακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια τις εκθέσεις μας και όπως είπατε τα δεδομένα μας είναι αξιόπιστα, συγκρίσιμα, ε, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ε, πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις και σκοπούς. Αλλά και για την, να αποφασίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι πιο συγκεκριμένα. Since you didn't, uh, there was no question δεν... About AGS δεν υπήρξε γι' αυτό ερώτημα, αλλά ήθελα πρώτα απ' όλα να μιλήσω για, τον, ε, για το Ινστιτούτο ως εργοδότη. Πρώτα απ' όλα, εγώ ως Διευθυντήρια, ως ε, ορίζους αρχή, πρέπει να υπογράψω κάτι συμβάσεις. Πρέπει, έχουμε υπογράψει λοιπόν συμβάσεις με 27 ανθρώπους, που είναι οι βασικοί υπάλληλοι, 27 και 28 κράτη-μέλη, 27 λοιπόν, να απλή πάλι, 10 συμβασιούχοι, που και αυτοί είναι μόνιμοι για το ΙΓΚΕ. Και μετά, εάν χρειαστεί να φύγει κάποιο με αδιαμετρότητα, με αναρωτική μακροχρόνια, έχουμε για κάποιου αναπληρωματικού που μπορεί να δουλεψει ενα ένα-δύο χρόνια, εξαρτάται πόσο του χρειαζόμαστε. Μετά έχουμε και του αποσπασμένου εθνικού εμπειρογνώμονε. Εδώ δεν υπάρχει σύμβαση, είναι δικοί του οι εργοδότε, ξεχωριστοί και δεν έχουμε κανένα, ε, καμία σύμβαση τύπου προσωρινού ή ε, διαλυπόμενη. Έχουμε, όπως είπατε και εσείς κυρία Μπλινκεβιτσιούτε, μέσω της συμφωνίας πλαισίου, της σύμβασης πλαισίου, έχουμε εταιρεία ε, προσλήψεων. Εκεί τα αναθέτουμε. Με διαφορετική λειτουργία. Ε, το βασικό που θέλω να είναι κατανοητό είναι ότι η οδηγία για τους προσωρινούς υπαλλήλους ερμηνεύεται και εφαρμόζεται λίγο διαφορετικά σε κάθε κράτος μέλος. Λόγω χαρή αυτό που βλέπουμε σε κάποιες χώρες, τους temporer τους μπερδεύουν ε, ως agent με τους workers, εργαζόμενοι ή υπάλληλοι. Για την ίδια θέση λέει η, Ευρωπαϊκή, η οδηγία ότι θα πρέπει ο μισθός να είναι συγκρίσιμος εάν ε, ο υπάλληλο έχει προσληφθεί για την ίδια θέση. Εμείς είμαστε συγκεκριμένη περίπτωση στην, ε, στο ΙΓΚΕ. Είμαστε πολύ μικρό Ινστιτούτο. Ίσως υπάρχει μια τεράστια διαφορά σε σχέση με τα μεγάλα Ινστιτούτα. Όλες οι τεχνικές διαδικασίες, προπολογισμό και το 27 συν 12 που έχουμε για υπαλληλικό προσωπικό δεν φτάνει Δηλαδή ακόμη και αν πάρουμε έναν ταμπορέρ, όπως είχαμε κάνει με τις συμβάσεις τις επόμενες, δεν μπορούμε να θέσουμε όσα μας λείπουν σε αυτόν τον συγκεκριμένο άτομο λόγω της ιδιαιτερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει δυνατότητα λοιπόν σύγκριση μεταξύ των interim και όσων απασχολούνται απευθείας από το ΕΓΚΕ. Έτσι κι αλλιώς οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες είναι διαφορετικές. Και όπω είπε η κυρία Μπλίνκεβιτ, ούτε το πρόβλημα ίσω να είναι ότι δεν έχουμε αρκετά για εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν είναι το πρόβλημα το χρήμα. Δεν είναι πρόβλημα ο ιδρυτικό κανονισμό. Η πρόταση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και δική σα σημαίνει ότι έχουμε μόνο 27. 27 υπαλλήλου. Ανθρώπου χρειαζόμαστε, όχι χρήμα. Δεν θα μα σώσει το χρήμα. Θέλουμε περισσότερο κόσμο. Κόσμο. Γιατί είμαστε πολύ μικροί Ευχαριστούμε για αυτές τις διευκρινήσεις. συζητήθηκαν και στα πλαίσια του προηγούμενων σημείων στην ημερήσια διαταξή. Τώρα ε, φτάνουμε στο τέλος της εξέτασης του σημείου αυτού. Απλώς να πω ότι όπως ξέρετε πρόσφατα εξελέγημεν τέλη Μαΐου. Όμως ως Επιτροπή ΦΑΜ ήδη είχαμε μια-δυο ευκαιρίες, φανταστικές ευκαιρίες να ενημερωθούμε για το ιστορικό, τη δουλειά σας, το τι κάνετε και έχουμε ωφεληθεί τρομερά από τη δουλειά του ΕΓΚΕ. Γι' αυτό λοιπόν μια τεράστια ευχαριστία για όλο το έργο σας, γιατί είσαστε πρωτοπόροι σε όλο αυτό το εγχείρημα και θέλουμε το ΕΓΚΕ να καταφέρει να ε, αποσπάει όλα αυτά τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για τις πολιτικές μας αρμοδιότητες. Θέλουμε να βασιζόμαστε σε στοιχεία, σε αξιόπιστες μεθόδους. Θέλουμε να αναπτυχθούν περαιτέρω Συγχαρητήρια λοιπόν για την δεκαετία δουλειά σα και κάθε τύχη και για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. So. we are coming to uh, uh, next point on the agenda. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Διακρίσεις με βάση ειδικά το φύλλο στα Δυτικά Βαλκάνια. Έχουμε καλέσει την κυρία Νικόλ Φάνσουερθ, διευθύντρια προγράμματος, ερευνήτρια στο κοσυφοπέδιο του δικτύου γυναικών συγκεκριμένα. Καλώς ήρθατε. Please, I invite Παρακαλώ, πάρτε το λόγο για την παρουσίασή σα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, μέλη του Κοινοβουλίου, για αυτή τη δυνατότητα. Είναι τιμή μου να μπορώ να παρακολουθώ τη δουλειά σα. Άκουσα και την παρουσίαση του ΕΓΚΕ και εμεί αντλούμε πολλά από τη δική του την έρευνα. Τώρα για τη δική μα την έρευνα θέλω να κάνω μια παρουσίαση για το δίκτυο γυναικών στο Κωσυφοπαίδιο. Έξι ενώ οργανώσει για την προστασία των γυναικών ε, στην Σουηδία. Προσθε... Χρηματοδοτούμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΣΥΝΤΑ για την καταπολέμηση τη ε, διακριτική μεταχείριση και τη ενισότητα στα Δυτικά Βαλκάνια. Εδώ υπάρχουν και κάποια φυλάδια τα οποία μπορείτε να πάρετε να τα διαβάσετε αν θέλετε, αλλά έχουμε και μεμονωμένε εκθέσει ανά χώρα, εάν σα ενδιαφέρει μια συγκεκριμένη χώρα. Η έκθεση αυτή είναι το εφαλτήριο γιατί έχουμε πολύ λίγα στοιχεία για την διάκριση βάσει των φύλων ε, και την ε, έμφυλη διάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε ως ακτιβιστές για να προσπιστούμε τα δικαιώματα. Εδώ υπάρχει μια ανάλυση, μια επισκόπηση, μελέτη με περισσότερες από 4.600 ε, συμμετέχοντες στα Δυτικά Βαλκάνια και αυτό γιατί ήταν ένα θέμα δύσκολο, ένα δύσκολο θέμα για να το θίξουμε και γι' αυτό ήταν ε, στο διαδίκτυο η μελέτη για να διατηρήσουμε την ανωνυμία των συμμετεχόντων. Αλλά βεβαίω εδώ υπάρχει και ένα ποσοστό σφάλματο στα ευρήματα. Διότι καταλαβαίνουμε ότι πολλέ φορέ έχουμε απαντήσει από ε, γυναίκε με εκπαίδευση που ζουν σε αστικά κέντρα και έχουν και κάποιο εισόδημα. Υπάρχουν λοιπόν πολλέ γυναίκε που έχουν πληγή από διακριτική μεταχείριση στην απασχόλησή του και Εδώ κάποια βασικά πορίσματα για τα θέματα μεταφοράς αφού μιλάμε για χώρες σε διαδικασία προσχώρηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και πού χρειάζεται ο ακτιβισμός, ε, οι κυβερνήσεις, τι βήματα πρέπει να κάνουν για να καταπολεμήσουν την ανισότητα. Είναι πολλές χώρες που έχουν πρόβλημα με τις εξαιρέσεις, δεν τις καταλαβαίνουν. Επίσης υπάρχει θέμα με το κατά πόσον ε, ε, όσοι έχουν πέσει θύματα δεν προστατεύονται στη συνέχεια αρκετά. Δεν υπάρχει προστασία για τις ε, αυτοαπασχολούμενες και βεβαίως και αντιστροφή του βάρους απόδειξης. μετά η σύσταση ενώσεων που θα μπορούσαν να προστατεύουν ε, τους, ε, τα θύματα διακριτικής μεταχείρισης, ούτε αυτές έχουν το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και μετά τα συζητήσατε και εσείς προηγουμένως για την εξισορρόπηση επαγγελματικού και γενικού σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης είναι ένα σημαντικό θέμα. Αδιαμητρότητας, πατρότητας, γονική, όλα προβληματικά σημεία και το νομικό πλαίσιο πρέπει να ε, συνάδει με την οδηγία. Ε, υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Επίσης, υπάρχουν θέματα υλοποίηση. Υπάρχει κατακαιρματισμό και στο νομικό πλαίσιο. Η διοικητική μεταχείριση καλύπτεται από διαφορετικού νόμου για την απασχόληση, την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση τη μεταχείριση και τον, ε, την εργασία, το εργατικό δίκαιο. Δεν είναι σαφέ ποιο ε, νομικό πλαίσιο που να χρησιμοποιείται κάθε φορά και υπάρχει σύγχυση. Τώρα, κάποιες από τις αντιλήψεις και τα ευρήματα από την έρευνα. Πρώτα απ' όλα τα ποσοστά απασχόληση στα Δυτικά Βαλκάνια. Βλέπετε σε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, σε όλε τι χώρε, να υπάρχει υψηλότερο ποσοστό απασχόληση για του άντρε από ότι για τι γυναίκε. Μακεδονία και Βοσνία και Ερσεγοβίνη. 19 ποσοστιαίε μονάδε η διαφορά στο χάσμα και 29 στο κοσφοπέδιο. Στο κοσφοπέδιο από όπου προέρχομαι, μόνο μία στις δέκα γυναίκες απασχολείται. Να το συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα της διάκρισης. Είστε παντρεμένες, έχετε παιδιά, έχετε χρόνο να έχετε παιδιά. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που θέτουμε στις περισσότερες γυναίκες σε συνεντεύξεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Και γενικώ ξέρουμε ότι οι εργοδότες ε, δεν προσλαμβάνουν γυναίκες λόγω της οικογένειας ή τη πρόθεση να έχουν οικογένεια. Πάνω από 50% των ερωτηθισών λένε ότι έχουν αντιμετωπίσει διακρίσεις στην πρόσληψή τους. Θα πρέπει βεβαίω να υπάρχει ε, πληρωμένη ε, μητρική άδεια. είναι και αυτό μια βασική πηγή διακριτική μεταχείριση για τι γυναίκε στην αγορά εργασία. Ε, γιατί δεν παίρνουν γονική άδεια γυναίκε επειδή του διακόπτουν τη σύμβαση, ε, άμεση αντίδραση ή εμέσω. Μειώνεται η σύμβασή του. Δεν θέλουν ε, ε, να συνεχιστεί η σύμβαση οι εργοδότε όταν είναι γυναίκε με γυναίκε. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με γυναίκε που έμειναν ανάγκε αφού έπιασαν δουλειά. Λένε το 1 πέμπτο ότι δεν πήραν καμία, αγωνική, καμία αμοιβή για την γονική τους άδεια, καμία απολαβή, ούτε από τον εργοδότη ούτε από την κυβέρνηση. Λέει μια γυναίκα, έχασα τη δουλειά μου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου, ενώ είχα μείνει τρία χρόνια στην εταιρεία και ε, με έδιωξαν μέσα σε μια εβδομάδα. 24 χρονών στη Βόρεια Μακεδονία. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι επίση διαδεδομένη στα Δυτικά Βαλκάνια. Κάθε μία στι τρει γυναίκε που έχει απαντήσει στην ε, στι συνεντεύξει μα, έχει υποφέρει από σεξουαλική παρενόχληση στην ε, δουλειά. Ο διευθυντή ήθελε να πλαγιάσει μαζί μου για να πάρω προαγωγή. Εδώ λοιπόν για την ε, διακριτική μεταχείριση βλέπουμε ότι πάνω από 76% όσοι είχαν πέσει θύματα, όσες μάλλον δεν το ε, κατήγγυλαν πουθενά και ένα άλλο ποσοστό, 4% πήγε στην αστυνομία, 3% έφτασε στα δικαστήρια και με νομική δίωξη και είναι πολύ λίγες αυτό που πέτυχαν κάποιο αποτέλεσμα. Δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου, γι' αυτό αντέχω και τα καταπίνω. Γυναίκα 47 ετών στο Μαυροβούνιο για όσου λοιπόν καταγγέλουν τη διακριτή μεταχείριση, οι περισσότεροι ήρθαν σε επαφή με του υπεύθυνου για την απασχόληση. Αλλά είναι πολλέ αυτέ που είπαν ότι και σε αυτή την περίπτωση έπεσαν θύματα έμφυλη βία. Τα πρόσφατα πορίσματα δείχνουν ότι περισσότερε άντρε και γυναίκε στα Δυτικά Βαλκάνια γνωρίζουν ότι τα θέματα στην εργασία που έχουν σχέση με το φύλλο είναι παράνομα, αλλά τα αντέχουν γιατί δεν ξέρουν, γιατί φοβούνται ότι αν τα καταγγείλουν θα είναι χειρότερα τα αντίπεινα μακροσκελείς δικαστικέ διαδικασίες, ε, καχυποψία για του δημοσίου θεσμού, να χάσουν τη δουλειά του τα έγγραφα δεν τα καταλαβαίνουν αυτά που αφορούν τη διακριτική μεταχείριση, τελικά δεν αποζητά κανεί ένδικη εκδίκαση τη υπόθεση. Η έρευνα αυτή βεβαίω κυρίω βασίζεται, όπω σα είπα, σε καλά εκπαιδευμένε ε, γυναίκε με δουλειά που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και ζουν σε αστικά κέντρα. Μία στι τρει όμω έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση παρόλα αυτά και πολλέ έμφυλοι ε, διακριτική μεταχείριση. Μπορείτε να φανταστείτε πώ είναι η ζωή για αυτέ τι γυναίκε που δεν βρισκόνται στην ίδια θέση με αυτέ που απάντησαν, που είναι σε ακόμα επισφαλέστερη θέση. Οι θεσμικές απαντήσεις ήταν ε, πολύ ισχνές. Λίγα στοιχεία τηρούν ε, οι θεσμοί και οι δημόσιες υπηρεσίες της χώρας μας. Βεβαίως αυτό δεν επιτρέπει να ε, βοηθήσουμε τον κόσμο που έχει πέσει θύμα εμφυλής βίας. Ε, βεβαίως τα θεσμικά όργανα δεν έχουν γνώση και εμπειρία, δεν έχουν ε, γνώση για την εμφυλή βία και τη διοικητική μεταχείριση και πώς πρέπει να αντιδράσουν σε τέτοιες περιπτώσεις οι δικές μας οι συστάσεις. Έχουμε κάμποσες, αλλά θα σας παρουσιάσω μόνο ορισμένες. Πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρξουν διορθώσεις στο νομικό πλαίσιο στα Δυτικά Βαλκάνια. Βλέπουμε τη διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως επίκαιρη και πολύ επικοδομητική για να προχωρήσουν αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται, ιδίω ό,τι αφορά για να βελτιωθεί η νομοθεσία μας βάσει τις οδηγίες της ίσης μεταχείρισης, τις οδηγίες των αυτοπροσχολουμένων και όπως είπα και προηγουμένω της εξορρόπησης επαγγελματικού και βίου. Είναι σημαντικά αυτά να βελτιώσουμε την εξισορρόπηση της εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας της χώρα μας. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε συστήσει ή μάλλον ασκείται πίεση για να υπάρξει θεσμική αναθεώρηση του συστήματος αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εργασιμότητα. Ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις και μέσα από τις αιτήσει ε, εκθέσεις αναχώρα και να ενθαρρύνει τα Δυτικά Βαλκάνια και τις κυβερνήσεις τους να βελτιώσουν το νομικό τους πλαίσιο βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών, κυρίως τις οδηγίες για την εξισορρόπηση επαγγελματικού και βίου. Επίση, νομίζουμε ότι υπάρχουν αρκετέ ευκαιρίε για την Ευρωπαϊκή Ένωση να το δει σε πολιτικό επίπεδο και να οργανώσει διάλογο για ζητήματα που αναφέρονται και στην έκθεσή μα για την αντιμετώπιση τη διακριτική μεταχείριση, τη διόρθωση του νομικού πλαισίου. Και είναι πολύ σημαντικό για μα, όποτε έρχονται βουλευτέ τη χώρα μα, να μιλούν και με ομάδε υπεράσπιση των γενικών των δικαιωμάτων, διότι αυτό προβάλλει και τη δουλειά μα. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει απευθεία, αλλά εμέσω. Είναι σημαντικό να δούμε και το νέο πουδουπού, το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, διότι εάν δούμε τον κοινό εφαρμοστικό κανονισμό, θα πρέπει να σκεφτούμε πώ η εξωτερική χρηματοδότηση μπορεί να ευθυγραμμίσει τη διάσταση ισότητα των φύλων. Αυτή τη στιγμή ο κανονισμό δεν έχει ξεκάθαρη πρόπτικη που να λαμβάνει υπόψη την ισότητα των φύλων. Είναι τελείω ασαφή. Εάν θέλουμε λοιπόν να πάμε στο κοινό εφαρμοστικό κανονισμό και να κοιτάξουμε την ευθυγράμμιση του βάση των φύλων, το κάναμε σε ένα έγγραφο που έτσι πειραματικά και θα το δείτε έξω την αίθουσα. Ε, εκεί βρίσκουμε πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να πιέσει όλου του δικαιούχου τη Ευρωπαϊκή ε, Χρηματοδότηση να λάβουν υπόψη την ισότητα των φίλων, ευθυγράμμιση. Επίση, πολύ ε, συγκεκριμένα υποχρεωτική υποβολή για την πρόοδο στο θέμα αυτό, βάσει των συστάσεων και του ΙΓΚΕ, του Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Και όπω είπε και η πρόεδρο προηγουμένω, ε, έχουμε και την ε, έκθεση Μούντι η οποία ζητούσε δείκτε συγκεκριμένου για τη διάσταση του φύλου που να χρησιμοποιούνται στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των δράσεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το πρόγραμμα δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όμω δεν είναι αρκετό το, ω προ του δείκτε. Δεν έχει ειδικού δείκτε και στοχευμένου. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν αυτέ οι προτάσει από το Κοινοβούλιο για να εφαρμοστούν. Έχουμε κάποιε ιδέε σε κάποια έντυπα για το πώ μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Τα βρείτε εκτό εθούση σε φυλάδια. Σα ευχαριστούμε τόσο πολύ για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Πραγματικά. Ε γνωρίζουμε το πρόβλημα στο χώρο εργασίας δεν είναι εύκολο στα Δυτικά Βαλκάνια και τελικά ποιοι υποφέρουν περισσότερο, πάντοτε οι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι θύματα της διακριτική μεταχείριση και όλων αυτών που αναφέρατε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για το link και θυμήσατε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής μας αυτά που ήδη γίνονται, ε, που έχουν κάνει και προηγούμενοι βουλευτές, η Μούντι για παράδειγμα, για το θέμα αυτό. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ξανά. Η κυρία Γιάροκα, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ξέρω το πεδίο έρευνά σα και θα ήθελα να πω κάτι για κάποια από τα ευρήματά σα και να σα μιλήσω για τι ε, δικές μας εμπειρίες στην Ανατολική Ευρώπη, γιατί τότε ε, είχαμε την ε, έκθεση Moody και υπήρχαν γυναίκες στην πρώην, ε, πρώην κομμουνιστικές χώρες, ε, των οποίων δεν γίνονταν σεβαστά τα δικαιώματα Πολλές ε, γυναίκες έχουν ήδη φύγει από τα Ανατολικά Βαλκάνια σήμερα και χάνεται έτσι ε, ανθρώπινο δυναμικό και μια ολόκληρη γενιά, διότι τελικά οι ηλικιωμένοι ε, δεν θα έχουν συντάξεις αν φεύγουν όλοι οι νέοι. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πολλούς διαφορετικούς τομείς και θα πρέπει αυτό το θέμα λοιπόν να το δούμε πιο σφαιρικά. Νομίζω λοιπόν ότι στα Δυτικά Βαλκάνια υπήρχε αυτή η στρατηγική για τους Ρωμά το 2011 και κάποιες στρατηγικές κατά της φτώχειας, αλλά αυτό που διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι τα πράγματα προχωράνε ε, αργά, πιο αργά από ό,τι στην Ανατολική Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν στα Δυτικά Βαλκάνια και χαίρομαι γιατί συμπεριλάβατε ένα τέτοιο ε, τμήμα στην ερευνά σας για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και να παρουσιάζονται κάποια εργαλεία για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Αν μου δίνετε λοιπόν λίγο περισσότερο χρόνο, θα ήθελα να πω στα θετικά ότι όχι μόνο στην εμπορία ανθρώπων, όπου υπάρχει ε, βεβαίως εδώ η υποχρέωση ικανοποίησης κάποιων κριτηρίων πριν την διαδικασία ένταξης. Αλλά θέλω να πω ότι πριν από κάποιες μέρες συναντήθηκα με τον συντονιστή κατά της εμπειρίας ανθρώπων και διαπίστωσα ότι υπάρχει πραγματική δέσμευση. Θα δοθεί λοιπόν συνέχεια στο θέμα. Ελπίζω λοιπόν ότι εδώ σε αυτή την Επιτροπή θα μπορέσουμε να σας στηρίξουμε όχι μόνο μέσω του PDP αλλά και των δικών μας προ ε, πρωτοβουλειών ε, ε, κατά κάθε είδους διάκρισης. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα, όχι μόνο εθνοτικά, αλλά υπάρχουν και προβλήματα στο κοψηφοπέδιο με παιδιά τα οποία ε, γεννιούνται με καρκίνο ή ε, κινδυνεύουν από ε, διάφορα μεταδιδόμενα νοσήματα και επίσης ότι δεν υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες ε, για να προσληφθούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Ναι, ε, θα πρέπει να γίνει λοιπόν αλλαγή πολύ γρήγορα σε αυτή την περιοχή. Το έργο σας θα βοηθήσει. Υπάρχει βέβαια το πρόβλημα πολλών φτωχών οικογενειών. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερο για την εκπαίδευση για ενημέρωση των γονέων ε, ε, και να έχουν και οι τοπικές κοινότητες καλύτερους ε, ηγέτες, καλύτερους επικεφαλής. Νομίζω ότι τα υφιστάμενα εργαλεία δεν τα χρησιμοποιούμε σωστά, διότι εσείς χρησιμοποιήσατε την κοινοτική οδηγία ΒΑΛ, αν όμω τα χρησιμοποιούσαμε αυτά τα εργαλεία, θα μπορούσαμε να λύσουμε πολύ περισσότερα προβλήματα. Διάκριση στο χώρο τη εργασία, για παράδειγμα. Αυτό το χρειαζόμαστε ιδιαίτερα. Αυτή η οδηγία θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να απαντήσετε. Ναι, χαίρομαι που θίξατε κάποια θέματα. Και θέματα λοιπόν που έχουν σχέση με τις διακρίσεις κατά των δύο φύλων. Η φροντίδα των παιδιών είναι από τα πολύ βασικά θέματα. Ε, το αναφέρατε και πριν. Ε, επίσης, τα διάφορα, διάφορες προκαταλήψεις στον χώρο εργασίας. Τώρα, όσον αφορά την ε, καλύτερη κατάρτιση του προϋπολογισμού και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ξεκινήσαμε να συζητάμε με προηγούμενα στελέχη της ε, Επιτροπής ΦΑΜ για το πώς θα μπορούσε να γίνει κάποια διάθεση κονδυλίων ε, που να έχουν να κάνουν ειδικά με ε, το θέμα της ισότητας των φύλων. Να υπάρχουν ειδικά κονδύλια και επίσης κονδύλια για την στέγαση και για την προσφορά υπηρεσιών για να μπορέσουν να προστατευθούν επίσης οι γυναίκες που έπεσαν θύμα βία. Ίσως λοιπόν να ε, διατεθούν ειδικά κονδύλια υπό το νέο PDP και να μπορέσουν οι γυναίκες έτσι να ε, λαμβάνουν περισσότερες υπηρεσίες. Βεβαίω όλα αυτά θα είναι και σύμφωνα με την σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Ελπίζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά θα συμβούν στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ήδη μας δώσατε μια ιδέα για το τι μένει να γίνει. Είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά στην Επιτροπή μας. Ε, πραγματικά συμβάλλατε με πολύ ανοιχτό πνεύμα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω. Ο Θεός είναι γυναίκα και το όνομά της είναι Πετρούνια. Αυτό είναι το φίλμ της ε, Βόρειας Μακεδονίας για το βραβείο Λουξ την περασμένη εβδομάδα. Ε, επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα σε θέματα τα οποία αναφέρατε ε, ήταν ένα πολύ ωραίο φιλμ. Αυτό για να ολοκληρώσω την παρουσίασή σας ε, με ένα θετικό στοιχείο, μια θετική προοπτική. Ευχαριστούμε πολύ. Και έτσι ολοκληρώνουμε. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα είναι στις 22 και στις 23 Ιανουαρίου του 2020 του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή σε όλους και ευχαριστούμε τους διερμηνείς.